Σα Σα ευχαριστώ πολύ. Well, thank you very much indeed, Minister. And we... Ευχαριστούμε, Υπουργέ, και εμεί ανυπομονούμε να συνεργαστούμε μαζί σα. Σημειώνουμε ότι οι γαλάζιες γραβάτες της Λιθουανικής Προεδρίας αλλά και νομβούλια θα είχαν προκαλέσει κάποια αναταραχή. Αλλά τέλος πάντων, εδώ είναι διαφορετικά τα πράγματα. Βλέπω την κυρία Στάιλερ εδώ που καταλαβαίνει τι εννοώ. Σας ευχαριστώ παντός για την δεξοδική και λεπτομερή παρουσίαση του έργου σας και που αναφερθήκατε και σε πολλές από τις εκθέσεις πρωτοβουλίας μας. Μας αρέσει να έχουμε την αντίδραση και την ανταπόκριση σε αυτές για να μπορούμε να προχωρήσουμε και να συνεχίσουμε το έργο μας και στην επόμενη θητεία. Σημειώνω αυτό που είπατε για τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς, κάτι που θα το επιδιώξουμε ενεργά ώστε να προχωρήσει και χαίρομαι πολύ που θέλετε να το προωθήσετε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξάμεινου. Αλλά υπάρχουν και άλλε εκθέσει ιδέα πρωτοβουλία, τι οποίε επεξεργαζόμαστε και η κυρία Γκέπχαρτ, η κυρία Μπίλτ, ο κύριο Γκυγιόν. Όλοι εργάζονται από αυτών των θεμάτων και σωστά από τις φοροτιμή στο έργο της κυρίας Πιτικάριαν και της κυρίας Αλντερμόζα. Θα έλεγα τώρα να ακούσουμε ερωτήσεις ε, ανά τρεις συναδέλφους. Έχουμε νομίζω άφθονο χρόνο για να μπορέσετε και να απαντήσετε. Και θα ήθελα να έχουμε ένα γύρο ερωτήσεων πρώτα από τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων. Η κυρία Φερχάιντα, η κυρία Γκέπχαρτ, ο κύριος Ζωσόρ, και η κυρία... Και η κυρία Ρούιλε. Α ακούσουμε την κυρία Φερχέιν, την κυρία Γκέπχαρτ και την κυρία Ρούιλε, ώστε να έχουμε τι τρει βασικέ ομάδε. Και αν θέλει και ο κύριο Ασφορτολόγο το λόγο μπορεί, αλλά α ακούσουμε πρώτα στις τρει κυρίε, Οι κυρίε προηγούνται. Äh, ευχαριστώ, Πρόεδρε, αξιότιμα Υπουργέ. Καταρχά, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για το γεγονό ότι ήρθατε εδώ πέρα και μα κάνετε μια παρουσίαση των προτεραιοτήτων σα. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό, θεωρώ. Και νομίζω είναι σωστό να συνεχιστεί το έργο που ξεκίνησε τα τελευταία ένα-δύο χρόνια. Και υπογραμμίζουμε να συνεχιστούν ακριβώ αυτέ οι δυο ε, Δύο-τρεις ερωτήσεις έχω να σας κάνω. Καταρχάς, ε, για την επικοινωνία σε ό,τι αφορά τη ε, βιομηχανική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εντοπίσει στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά και νέα καινοτόμα φαρμακευτικά προϊόντα μας καθιστούν πραγματικά απαραίτητη την, κατάσταση μιας στρατηγικής σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα, την διαθεσιμότητα πολύ σημαντικών φαρμακευτικών προϊόντων, αλλά και σε ό,τι αφορά την διατήρηση της, ε, των εργοστασίων εδώ στην Ευρώπη. Και τα καινοτομικά αυτά φαρμακευτικά προϊόντα είναι πάρα πολύ σημαντικά για την Ευρώπη και μας ανησυχεί ιδιαίτερα το γεγονός αυτό ως πολιτική και στην Επιτροπή αλλά και στο Κοινοβούλιο. Και οι περικοπές σε κάποια κρατή-μέλη λόγω της κρίσης αποτελούν μεγάλο πρόβλημα. Και εδώ η Λιθουανική Προεδρία θα πρέπει να κάνει μια σχετική συζήτηση. Ένα δεύτερο ερώτημα. Είπατε κι εσείς ότι η ψηφιακή ατζέντα και η προτεραιότητα για μέτρα ενίσχυση της αξιοπιστίας της ψηφιακής αγοράς θα αποτελέσει η προτεραιότητά σας. Η κυρία Κρούς, σε μία από τις τελευταίες συνδυάσεις που είχαμε μαζί της, εξήγηλε ένα αρκετά εκτεταμένο πακέτο σε ό,τι αφορά τον τομέα των τηλεπικοινωνιών, σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την κατάργηση των τελών ε, περιαγωγής Για τη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς στον τομέα των τηλεπικοινωνιών γιατί η αγορά αυτή είναι πάρα πολύ κατακρεματισμένη σήμερα. Και τώρα λοιπόν σας ερωτώ ποια είναι η δική σας στάση. Υποστηρίζετε ως Λιθουανική Προεδρία αυτές τις πλειοδοξίες. Uh, σας ευχαριστώ κύριε Γεπχάρτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, καλώς ορίσατε καταρχάς. Είσαστε η πρώτη Προεδρία νομίζω από τα κράτη της Βαλτικής. Είναι μια μεγάλη πρόκληση αυτή για εσάς. Θα δώσετε νέα, αν θέλετε, διάσταση σε αυτό το έργο. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μαζί μπορούμε να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Μιλήσατε για κάποια πολύ σημαντικά θέματα. Καταρχάς, η οδηγία για υπηρεσίε και η εφαρμογή της. Αυτό ασφαλώς μας απασχολεί ιδιαίτερα εδώ στο Κοινοβούλιο. Έχουμε δουλέψει σκληρά προς την κατεύθυνση αυτή. Και φυσικά θέλουμε να είναι σωστή και η εφαρμογή. Είπατε ότι ελπίζετε να σας υποστηρίξουμε σε κάθε περίπτωση. Θα σας υποστηρίξουμε ιδιαίτερα από την ομάδα μου. Θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι μια ένωση των πολιτών, με ανοιχτή αγορά, στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Υπάρχουν λοιπόν τρία ζητήματα τα οποία θα συζητηθούν τον επόμενο καιρό και τα οποία άπτονται ιδιαιτέρως της προστασίας του καταναλωτή. Ένα το αναφέρεται ήδη για τα εργοστάσια παραγωγής, ηλεκτροπαραγωγής. Έλαβα τρεις επιστολές μόλις τις τελευταίες ημέρες από πολίτες που έχουν προβλήματα. Ένας πατέρας, για παράδειγμα, Συγγνώμη, μεταφορά των οχημάτων. οχημάτων. Ένα πατέρα ο οποίο πήρε ένα αυτοκίνητο για την κόρη του η οποία παντρεύτηκε και δεν μπορεί να το εξάγει στην χώρα που τυχαίνει να ζει η κόρη του. Είναι σημαντικά ζητήματα αυτά. Ένα άλλο δεύτερο θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό για του πολίτε είναι το θέμα του roaming, τη περιεγωγή. Σα ρώτησε, συνάδελφο ποια είναι η δική σας ε, στάση. Είναι γεγονός ότι στην μεγάλη ενιαία αγορά που έχουμε δεν είναι δυνατόν να χρεώνονται τέλη περιαγωγή. Και μεταξύ Κιέλου και Στρασβούργου να υπάρχουν διαφορές στην τιμολόγηση. Δεν είναι δυνατόν να εξακολουθούν να υπάρχουν τέτοιες διαφορές στις τιμές. Πείτε μας λοιπόν τη δική σας στάση. Τρίτο και τελευταίο θέμα το οποίο θέλω να αναφέρω. Οι βασικοί λογαριασμοί. Και αυτό με απασχολεί ιδιαίτερος. Ο κύριος Μπαρνιέ πρότεινε ένα νομοθετικό πακέτο και θα ήθελα λοιπόν και εσείς να μας πείτε ποια είναι η στάση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ξέρω, στη δική μου χώρα ότι δεν ε, συμφωνούν μαζί μου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσω να προασπίζω την άποψή μου αυτή για το θέμα αυτό. Θέλουμε οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε τέτοιους βασικούς λογαριασμούς. Γιατί δάλλως δεν μπορεί κανείς να συμμετέχει πραγματικά στην κοινωνία, χωρίς λογαριασμό δηλαδή. Uh, κυρία ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Χαίρομαι ιδιαίτερα που θα συνεργαστούμε μαζί. Θεωρώ ότι θα είναι φιλόδοξη και πολύ σημαντική η συνεργασία αυτή, γιατί εξακολουθεί να μένει ανοιχτό ένα πολύ μεγάλο νομοθετικό πακέτο. Η κυρία Σάλτεμου μίλησε για την ασφάλεια των προϊόντων, για την επιτήρηση και την υποπτήρια τη αγορά. Και το είναι ερώτημα το κατά πόσο θα τα περάσουμε αυτά μέσα στην τρέχουσα θητεία γιατί με την κυρία Σάλντε Μούζα ε, συμμετείχα και σε ό,τι αφορά το πακέτο για τα αγαθά και αυτό πήρε πάρα πολύ χρόνο. Γι' αυτό λοιπόν ε, επιθυμώ να σημειωθεί πρόοδος. Ύστερα, μία άλλη ιδιαίτερα επιθυμία η συνάδελφός μου, η κυρία Ρόιτοβα, εδώ και πολλά χρόνια έχει πρόβλημα με το alignment package. Θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό εάν θα μπορούσατε εσείς να κλείσετε το πακέτο αυτό προκειμένου και να ψηφιστεί στη συνέχεια, γιατί είναι, ξέρετε, πάρα πολύ σημαντικό μετά από τόση συζήτηση και τόση δουλειά να έχει ο τέλος το πακέτο αυτό και φυσικά αυτό είναι από σε τελική ανάλυση στο Συμβούλιο. Ο κύριος Υπουργό. Θέλετε να απαντήσετε στις ερωτήσεις αυτές, στις τρεις αυτές ερωτήσεις και στη συνέχεια θα έχουμε άλλο ένα γύρο ερωτήσεων. Η κυρία Βερνιό, η κυρία Ράπτη και η κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κατά πρώτον, να σας ευχαριστήσω για τις ε, ευχές σας και τη στήριξη για το πρόγραμμα εργασιών μας. Πραγματικά εργαστήκαμε σκληρά για να το καταρτήσουμε και σας είμαστε ευγνώμονες. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους συντονιστές της Επιτροπής σας που μόλις πήραν το λόγο και είπαν ότι όσα έχουμε κάνει οι προθέσεις δηλαδή που έχουμε δείξει είναι, εκτιμώνται. Και εμείς βεβαίως εκτιμούμε το δικό σας έργο. Σε ό,τι αφορά τις ερωτήσεις αυτές καθ' Κατά πρώτον, για την κυρία Φαρχέιν. Ρώτησε τι γίνεται με την φαρμακοβιομηχανία και τα σχετικά ζητήματα. Όντως, είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Εάν κοιτάζετε το πρόγραμμά μας, θα καταλαβαίνετε πόση έμφαση έχουμε δώσει στην ανταγωνιστικότητα και οτιδήποτε σχετίζεται με αυτή. Για μας αποτελεί προτεραιότητα της Προεδρίας μας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν το έργο μας με το άτυπο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας τον Ιούλιο στο Βίλνιους και τον Σεπτέμβριο σκοπεύουμε να διοργανώσουμε συζήτηση όπου ελπίζουμε να υπάρξει συμμετοχή και έντονη στρίξη και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τον Σεπτέμβριο θα αξιολογήσουμε όλες τις προτάσεις, όλες τις ιδέες που θα ακουστούν, ώστε να πηχηθούν στα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την σχετική πολιτική. Ελπίζουμε ότι τα συμπεράσματα αυτά θα χρησιμεύσουν ως βάση και θεμέλιο για το 2014 για το Συμβούλιο του Φεβρουαρίου συγκεκριμένα. Η επόμενη ερώτηση είχε να κάνει με τις ε, προτεραιότητές μας για την ψηφιακή ατζέντα. Ήδη ανέφερα στην παρουσίασή μου ότι αυτή είναι μία από τις προτεραιότητές μας. Θέλουμε να εφαρμόσουμε την ψηφιακή ατζέντα για την εσωτερική αγορά στο δυνατόν συντομότερα, για να αρχίσει να λειτουργεί εύρυθμα. Γι' αυτό έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Για πιο συγκεκριμένα μέτρα, να αναφέρω με παραδείγματα κάποιους τομείς για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις ε, προστατευμένες υπηρεσίες. Θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ευρωκοινοβούλιο εδώ και θα προσπαθήσουμε επίσης να επιτελέσουμε πρόοδο και στις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές τηλεπικοινωνίες. Ελπίζουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία και να έχουμε την στήριξη του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή τουλάχιστον να εκκινηθούν οι συζητήσεις και οι συνομιλίες με το Ευρωκοινοβούλιο. Θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε και στο δίκτυο πληροφοριών καθώς και τη σχετική ασφάλεια και την οδηγία που τα αφορά. Επίσης ε, για το ευρυζωνικό διαδίκτυο θα το συζητήσουμε και αυτό και θα προσπαθήσουμε να το προχωρήσουμε. Thank ε, Γκέπχαρντ. Για την κυρία Γκέπχαρντ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις προτάσεις σας και για την προθυμία σας να συνεργαστούμε. Το εκτιμώ ιδιαίτερος. για την εγγραφή οχημάτων. Κατά την Ιρλανδική Προεδρία υπήρχαν πολλά σχόλια από τα κράτη-μέλη για αυτή τη συγκεκριμένη νομική πράξη. Μίνιστρο, ε, Εδώ μας απασχόλησε αυτό σε επίπεδο Συμβουλίου Υπουργών Ανταγωνιστικότητας και όπως ε, και η Κύπρος και η Ιρλανδία θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε το θέμα αυτό ώστε να επιταχυνθούν οι σχετικέ διαδικασίε και να περιοριστεί το διοικητικό άχθο, διότι πραγματικά αποτελεί φραγμό για την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών. Θέλουμε να έχουμε πραγματικά μια ισχυρή εντολή για τι σχετικέ διαπραγματεύσει. Το άλλο σας ερώτημα είχε να κάνει με τους βασικούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Και αυτό σχετίζεται με την ψηφιακή μας ε, ατζέντα και όπως ε, υπονόησα θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια και προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να επιτύχουμε μια συμφωνία. Κυρία Ρίλε, θα προσπαθήσω να απαντήσω και στα δικά σας ερωτήματα τώρα. Για την ασφάλεια των προϊόντων και τη σχετική δεσμευμέτρων. μέτρων. Είναι πραγματικά ένα θέμα σοβαρό, όπως και η επαγρύπνηση, η παρακολούθηση της εσωτερικής αγοράς. Τα δύο αυτά ζητήματα είναι αλληλένδετα και στόχος μας είναι να επιτύχουμε πρόοδο και εδώ. Θέλουμε η πρόοδος αυτή να είναι ορατή, να φανεί η δουλειά μας δηλαδή. Είναι μία προτεραιότητα γιατί συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο για την εσωτερική αγορά, το δεύτερο πακέτο και θα πρέπει να συμπληρωθεί και από νέε πρωτοβουλίε. Θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε ισορροπία μεταξύ την ασφάλεια των προϊόντων και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Βεβαίως, ε, αυτή η πρόθεση σημαίνει ότι θα πρέπει να αναλάβουμε σοβαρή δράση και αυτό σκοπεύουμε και να κάνουμε. Έχω μελετήσει τις σχετικές προτάσεις και πραγματικά θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με το Ευρωκοινοβούλιο γιατί χρειαζόμαστε την στήριξή σας για να προχωρήσουμε. Θα υπολογίζουμε στην συνεργασία της κυρίας Πιτικάινεν και της κυρίας Σαλντεμόζε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στις σχετικές διαπραγματεύσεις. Ελπίσεις, ελπίζουμε ότι το Νοέμβριο θα ξεκινήσει η φάση των τριμερών διαλόγων. Σας ευχαριστώ. Eh, Για το δεύτερο ερώτημά σας. Για την ευθυγράμμιση με τις απαιτήσεις του νέου συστήματος. Στα τελευταία στάδια των δημοτεύσεων είχαμε κάποιες δυσκολίες. Και αυτό είχε αρκετές συνέπειες οριζόντιου χαρακτήρα σε όλες τις νομοθετικές προτάσεις που σχετίζονταν με, αυτή τη, με αυτές τις διαπραγματεύσεις. Δεν ολοκληρώθηκε λοιπόν η εκδοχή της πρότασης εντός Ιρλανδικής Προεδρίας, αλλά πιστεύουμε ότι επί Λιθουανικής Προεδρίας θα καταβάλουν όλοι κάθε δυνατή προσπάθεια για να προχωρήσουμε και να καταλήξουμε σε συμφωνία. Ευχαριστώ. Ωραία. Σας ευχαριστούμε. Δεν ξέρω αν το αναφέρατε συγκεκριμένα, αλλά από τη θέση μου ως Πρόεδρο για την πρόταση περιαγωγής που αφορά το έργο της κυρίας Κρούς δεν είναι μόνο θέμα δικής μας αρμοδιότητας, αλλά πάντοτε έχουμε εδώ πολύ ισχυρέ απόψεις και συζητούμε με την κυρία Κρούς και για τη διάσταση που αφορά τα δικαιώματα των καταναλωτών, οπότε και εμάς μας είναι προσφυλές το θέμα αυτό. Να ακούσουμε την επόμενη σειρά ομιλητών, η κυρία Βερνιό, η κυρία Ράπτη και η κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Η κυρία Βερνιό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε που ήρθατε τόσο γρήγορα για να μας παρουσιάσετε το πρόγραμμα της Λιθουανικής Προεδρίας και τη προτεραιότητά σα για τα θέματα εσωτερική αγορά και προστασία των καταναλωτών. Συχνά παραθέτω τον Ζακ Ντελόρ και είναι φυσικό για τη μεγαλίδα. Ο Ζακ Ντελόρ έλεγε να μην ερωτευτούμε την εσωτερική αγορά και έχει δίκιο. Είχε δίκιο γιατί ε, η πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η βάση της ανταγωνιστικότητάς μας. Χάρη σε αυτές μπορούμε να, να έχουμε ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Αλλά δεν ιδιοποιούμαστε σωστά την εσωτερική αγορά, δεν την αφομοιώνουμε σωστά. Οι καλύτεροι νόμοι πολλές φορές μεταφέρονται κατά τρόπο εσφαλμένο. Υπάρχουν πολλές φορές δυσκολίες αναφέρατε την οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα και σα ευχαριστώ γιατί νομίζω ότι όντω και με την Ελληνική Προεδρία εργαστήκαμε πολύ αποτελεσματικά για το θέμα αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να μα πείτε ποιο θα είναι αντίκτυπο τις οδηγίες για τι υπηρεσίε, τι πιστεύετε ότι θα γίνει και τι θα γίνει με, τι θα γίνει με την ε, αναγνώριση των ε, των των πολιτών η κινητικότητα είναι πολύ σημαντικό, σημαντικό στοιχείο για τους πολίτες και να σας πω ότι στη χώρα μου τα πράγματα δεν πάνε καλά και η Γαλλία είναι από τις τρίτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρεται επίσης την εσωτερική αγορά και το τι γίνεται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτό σχετίζεται και με τι προτάσει του κυρίου Μπαρνιά για τι τραπεζικέ υπηρεσίε. Πιστεύετε ότι θα μπορέσετε σύντομα να παρουσιάσετε ένα κείμενο, να το, να το υποβάλλετε για να τελειώσει αυτό το χάο και να υπάρξει επιτέλους διαφάνεια για τους τραπεζικούς ε, δασμούς ε, και τις προμήθειες εντός ε, μιας και μόνης χώρας, γιατί μεταξύ τραπεζών πολλές φορές υπάρχουν μεγάλες διαφορές, αλλά και μεταξύ των χωρών όλων. Είναι θέμα εσωτερική αγοράς και αυτό. Και έπειτα τι σκοπεύετε να κάνετε με την ανάγκη να συνεργαστούμε πραγματικά για τις καθυστερήσεις πληρωμών. Εδώ πρέπει κάτι να γίνει με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πολλές φορές αναγκάζονται να κατεβάσουν ρολά διότι τα τιμολόγια τους δεν καλύπτονται συστηματικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Μπερναντέτ. Η κυρία Ράπτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, να ευχαριστήσω πρώτα τον κύριο Υπουργό γιατί στην εισήγησή του αναφέρθηκε και στο θέμα των τελωνίων και στο θέμα των υπηρεσιών ε, είχα την χαρά και την τιμή να εργαστώ μαζί με την κυρία Λεγκρίπ ως σκιώδης εισηγήτρια για το θέμα της αναθεώρησης του Τελωνιακού Κώδικα, όπως επίσης είχα την χαρά και την τιμή να συνεργαστώ με την κυρία Κοράτσα Μπίλτα για το θέμα των υπηρεσιών. Άρα από την εισήγησή σας, με την εισήγησή σας, μου αφαιρέσατε δύο ερωτήσεις που είχα να κάνω. Περνάω λοιπόν στην τρίτη ερώτηση κατευθείαν που έχει να κάνει με ένα θέμα που αγγίζει νομίζω όλες τις δραστηριότητες της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς. Η συνθήκη της Λισαβόνας, όπως ξέρετε και ξέρουμε όλοι μας, στο άρθρο 9 λέει πάρα πολύ απλά ότι καλούμαστε να λαμβάνουμε υπόψη μας όταν χαράζουμε τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ε, δημιουργία από τη μια πλευρά υψηλού επίπεδου απασχόλησης και από την άλλη μεριά τη διασφάλιση της κοινωνικής προστασίας των Ευρωπαίων πολιτών. Με άλλα λόγια, σε κάθε κίνηση που αφορά την οικονομική ανάπτυξη πρέπει να έχουμε υπόψη μας τις κοινωνικές επιπτώσεις. Διαβάζοντας το πρόγραμμα της Προεδρίας είδαμε πολύ χαρά ότι πάντα η προτεραιότητα δίνεται με μια ισορροπία. Από τη μια μεριά οικονομική ανάπτυξη, από την άλλη μεριά κοινωνική προστασία και ασφάλεια. Και ρωτώ ευθέως κύριε Υπουργέ, είστε έτοιμοι ως Λιθουανική Προεδρία να προωθήσετε, να ζητήσετε, να εισηγηθείτε την κοινή συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών με τους, υπουργό, με τους Υπουργούς των Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της κοινωνικής διάστασης. Ευχαριστώ. Thank you very much. And finally in this round, Mrs. Ευχαριστούμε. Και τελευταία στο γύρο αυτό, η κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Θέλω και εγώ να καλωσορίσω θερμά τον Υπουργό και την Προεδρία σας. Πραγματικά χαίρομαι που ανελαμβάνει μια βαλτική χώρα, μια χώρα της Βαλτικής δηλαδή, γιατί υπολογίζω πολύ στην συνεργασία σας. Ευχαριστούμε λοιπόν για την ενημέρωση και που μεταφέρατε σωστά και προωθήσατε την οδηγία για την ψηφιακή αγορά και που την προωθείτε, την οδηγία επίση για τι υπηρεσίε. Έχουμε την ευθύνη να δημιουργήσουμε θέσει εργασία στην Ευρώπη και να τονώσουμε την απασχόληση. Είμαι τώρα υπεύθυνη για μια έκθεση μεταξύ των οποίων οι συνάδελφοι, η κυρία Γκέμπχαρτ, ε, έχουν, ο κύριο Χάρμπορ έχουμε επιτελέσει εξαιρετικό έργο. Και θέλουμε πραγματικά να δείξουμε στο Συμβούλιο ότι πρέπει αυτό να περιληφθεί ως πρώτη προτεραιότητα στην, στον κατάλογο προτεραιοτήτων του Συμβουλίου και να μείνει και στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας ε, και στο Συμβούλιο για την Ιστορική Αγορά ως ένα από τα πρώτα θέματα. Στερούμε θέσεις εργασίας από τον κόσμο, τη στιγμή που δεν υπάρχουν κονδύλια του κράτους και δεν υπάρχουν κίνητρα. Έτσι λοιπόν δεν λέω ότι θέλουμε να επιβάλλουμε κάτι, αλλά πραγματικά μόνο να ακούσω και τι απόψει σας για συγκεκριμένα ζητήματα. Τα άρθρα 15 και 17. Οι ε, ε, λόγοι δημόσιου συμφέροντο θα θέλαμε το Συμβούλιο να τερμινεύσει αυτά περισσότερο αναλογικά, ιδίω από την πλευρά κάποιων κρατομελών, να μην χρησιμοποιούνται για να μπουν από το παράθυρο ε, περιορισμοί που ουσιαστικά μεταφράζονται σε προστατευτισμό. Τα θέματα τη προστασία καταναλωτών, ε, κάποιοι περιορισμοί. Δεν είναι δικαιολογημένα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξέρει ότι ετοιμάζει μια αναφορά για το Συμβούλιο και να δείξει τη δική της προσέγγιση για τη μεγιστοποίηση των, ε, οικονομικών, ε, των ωφέλιμων οικονομικών συνεπειών. Αυτό είναι πολύ καλή ιδέα, αλλά υπάρχουν κάποια κάτι μέλη τα οποία αρχίζουν και γίνονται ανυπόμονα και θέλουν την ενισχυμένη συνεργασία και να προχωρήσει έτσι το θέμα. Εγώ δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ διότι δεν είναι η στιγμή να υπάρξει κατακαιρματισμό στην εσωτερική αγορά. Υπάρχει ανάγκη να δείξουμε ότι μπορούμε να υλοποιήσουμε το 28 πολύ γρήγορα και να φανούν χειροπιαστά αποτελέσματα. Ελπίζω ότι και εσείς αυτό το στόχο θα επιδιώξετε. Ψηφίζουμε αύριο στην Επιτροπή μας για την Οδηγία των Υπηρεσιών και ελπίζω ότι θα υπάρξει πραγματικά μια μαζική πλειοψηφία μετά την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε με την κυρία Ρίλο, την κυρία Ράπτη και όλους τους άλλους συζητητές και τον κύριο Χάρμπορ. Ελπίζω κύριε Χάρμπορ πραγματικά να μπορέσουμε να παραμείνουμε πιστοί στο στόχο που έχουμε θέσει και να περάσει αυτό το μήνυμα στο Συμβούλιο. Επίσης θα ήθελα να σας καλέσω να σκεφτείτε στις προτεραιότητές σας, να σκεφτείτε και τον τομέα των λιανικών ελληνικών πωλήσεων, της ελληνικής αγοράς. Εργάζομαι χρόνια στο Ευρωκοινοβούλιο και έχουν κάνει κι άλλοι εξαιρετική δουλειά για το θέμα αυτό, αλλά πραγματικά είναι πολύ καλός τρόπος για να υπάρξουν περισσότερες θέσεις εργασίας. Χρειαζόμαστε έναν πιο αποτελεσματικό, πιο βιώσιμο και πιο δίκαιο τομέα λιανικής αγοράς. Υπάρχουν ε, πολλές ε, εθελοντικές πρωτοβουλίες, πολλές ε, προσπάθειες αυτορύθμισης και έχουμε δει τα αποτελέσματα στις Βρυξέλλες. Πρέπει να αναλάβουν ευθύνες στα κράτη-μέλη και να έρθουν πιο κοντά εταιρείε λιανικής τους πολιτές, τους αγοραστές δηλαδή. Ε, πρέπει αυτή την αρμοδιότητα να την αναλάβει το Συμβούλιο να τη φέρει εις πέρας. Σας ευχαριστώ. Ωραία. Ευχαριστούμε. Πολλές ερωτήσεις και κάτι τελευταίο. Ίσως καθυστερήσατε, αλλά να πω ότι η Λιθουανική Προεδρία είπε ότι θα στηρίξει μέτρα για την λιανική αγορά και για να ενθαρρύνει και τις σχετικές εργασίες της ομάδας υψηλού επίπεδου. Είμαι βέβαιος ότι ο Υπουργός θα συμπληρώσει την προηγούμενη παρατηρήσή του, αλλά απλώ να σας το ξεκαθαρίσω γιατί το είπε στην ανακτήρια ομιλία του. Υπουργέ, έχετε το λόγο για να απαντήσετε σε αυτούς τους τρεις ερωτώντες. Και μετά έχουμε την κυρία Στάιλα και την κυρία Σάλντε Μόζε στον επόμενο γύρο ομιλητών και οποιοδήποτε άλλο δεν έχει πάρει ως τώρα το λόγο μπορεί να το ζητήσει. Μπορεί να προλάβουμε και δεύτερο πάνελ. Ας ακούσουμε πρώτα αυτές τις ερωτήσεις. Πρόεδρε, κατά πρώτον, θα απαντήσω στις ερωτήσεις της κυρίας Βερνιώ. Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις σας ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις όντως περνούν δύσκολες στιγμές. Θα πρέπει κάποιες φορές οι οδηγίες να μεταφέρονται με μεγαλύτερη προσοχή και να μην γίνονται σφάλματα. Προσπαθούμε λοιπόν να επιστήσουμε την προσοχή των κρατών και να τα ενθαρρύνουμε ώστε να ξαναδούν την νομοθεσία της εσωτερικής αγοράς, να διορθώσουν αυτά που δεν πάνε καλά και να τα μεταφέρουν σωστότερα. Σε ό,τι φορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το όντι. Θα αναλύσουμε το πώς έχει μεταφερθεί η οδηγία για τις μικρές επιχειρήσεις σε μια από τις συνόδους του Συμβουλίου και θα είναι και ένα από τα θέματα ενός από τα άτυπα συμβούλια που πρόκειται να ε, διεξαχθούν τον, τον Ιούλιο. Θέλουμε να δούμε όλες τις ε, πρωτοβουλίες που θα τονώσουν τις μικρές επιχειρήσεις, το Think Small δηλαδή. Όσο για την οδηγία για τα ε, ε, επαγγελματικά προσόντα. Οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων, μάλλον συγγνώμη, η οδηγία για τις καθυστερημένες πληρωμές. Ε, πολλές ε, επιχειρήσεις έχουν υποβάλει παράπονα και προσφυγές για το θέμα αυτό και θα πρέπει μαζί με την πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις να το δούμε αυτό με ιδιαίτερη προσοχή στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας. Μετά, για τις τραπεζικές υπηρεσίες. Να σας πω το εξής. Πριν έρθω στην σημερινή συνάντησή μας, συνάντησα τον Υπουργό Οικονομίας, διότι το θέμα αυτό έπιπτε στο δικό του πεδίο αρμοδιότητων και επιβεβαίωσε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να επιτευχθεί πρόοδος σε αυτό το τομέα. ράπτε, Τώρα, για τις ερωτήσεις της κυρίας Ράπτη. Μου θέσατε διαφορετικές ερωτήσεις κι εσείς και για, τα, για τις τελωνιακές ε, υπηρεσίες, για την οδηγία των υπηρεσιών. Συμφωνώ με την παρατηρήσή σας εδώ ότι χρειάζεται η σωστή ισορροπία μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης, της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και των κοινωνικών προοπτικών. Όλα τα θέματα αυτά είναι αλληλένδετα και θα πρέπει να συμβαδίζουν. Δεν πρόκειται η οικονομία να αναπτυχθεί εάν δεν υπάρξουν νέε θέσει εργασία και αν δεν προστατεύσουμε και τα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων. Ρωτήσατε εάν αυτή την αρχή θα τη σεβαστούμε. Αναμφίβολα και αναντήρητα θα την ακολουθήσουμε πιστά. Ήδη ανέφερα ότι μια από τις προτεραιότητές μας είναι η ασφάλεια των προϊόντων και η παρακολούθηση της εσωτερικής αγοράς και το σχετικό πακέτο, η δέσμη μέτρων. Θα φροντίσουμε να βρούμε την σωστή ισορροπία μεταξύ των δύο αυτών στοιχείων, της ασφάλειας των προϊόντων και της παρακολούθησης της εσωτερικής αγοράς. Όσο για την κυρία Κοράτσα Μπίλτ και τις δικές της ερωτήσεις για την ε, λιανική αγορά, το λιανεμπόριο. Βεβαίως και αποτελεί μέρος των προτεραιοτήτων μας. Και θα τα εξετάσουμε τα ζητήματα αυτά και θα τα προωθήσουμε. Θα προσπαθήσουμε μέχρι το 2014 να εγκρίνουμε το πρόγραμμα για τους καταναλωτές 2014-2020. Και σε ό,τι αφορά την οδηγία για τις υπηρεσίες. Θα είμαστε ευγνώμονες στο Ευρωκοινοβούλιο εφόσον μας έστελνε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις του σχετικά. Πραγματικά αναμένουμε την συνεισφορά σας στο τομέα αυτό και για την οδηγία των υπηρεσιών συγκεκριμένα η αρχική ημερομηνία υλοποίηση ήταν το 2009. Έπρεπε ω τότε η οδηγία να έχει μεταφερθεί σωστά. Ωστόσο, γνωρίζουμε σήμερα ότι το ΑΕΠ ε, αυξανόταν κατά 0,8% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το δυναμικό που θα έπρεπε να έχουμε αντλήσει από την ε, πρόταση αυτή δεν έχει δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώ. Θα πρέπει να έχουμε αύξηση του ΑΕΠ κατά 2%. Οπότε, βεβαίω ακόμη έχουμε τεράστιε δυνατότητε. Η μεταφορά τη οδηγία των υπηρεσιών λοιπόν είναι κάτι που θα μα απασχολήσει και θα φροντίσουμε να δούμε και τα σχετικά ζητήματα όπως ε, τα νομικά προβλήματα, τη σωστή υλοποίηση της οδηγίας και το πώς θα αξιοποιήσουμε καλύτερα τα ενιαία σημεία επαφή. Το ανέφερα στο Συμβούλιο ανταγωνιστικότητα και θα κοιτάξουμε το Δεκέμβριο να ετοιμαστούν συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ε, πολιτική της ε, εσωτερικής αγοράς. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου να απεικονίζουν και την ανασύσταση χώρες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου της, αναχώρασης τάσης συγγνώμη, του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Και επίσης, σας διαβεβαιώ ότι θα δούμε πολύ συγκεκριμένα κάποιους περιορισμούς που ήδη γνωρίζουμε επειδή το έχουν επισημάνει επιχειρήσεις στη Λιθουανία και τα θέματα αυτά θα συζητηθούν και στα ε, άτυπα και στα επίσημα ε, Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητα. Θα αναφέρουμε το τι γνωρίζουμε εμεί από τη δική μα χώρα, με τα δικά μα παραδείγματα και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συζητηθεί το θέμα αυτό όσο πιο διεξοδικά γίνεται. Αυτά θα μπορούσα να σα απαντήσω προ τη στιγμή. Ευχαριστώ. Good. Uh, thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Τέλερ Σαρλεμόσα, ο Σβάμπ μήπως, δεν ξέρω αν θέλετε κι εσείς να ρωτήσετε κάτι συζητήσαμε την διακυβέρνηση της ενίας αγοράς. Το συζητήσαμε πριν. Ο Λιθονός, ο Υπουργός το έχει βάλει το θέμα αυτό σαν μία από τις πρώτες προτεραιότητές του. Αν ε, θέλετε λοιπόν κάτι να ρωτήσετε σχετικά, έχουμε χρόνο. Παρακαλώ λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κύριε Στήλε, ευχαριστώ και τον Υπουργό που ήρθε σήμερα. Θέλω να προσθέσω δύο πράγματα στα όσα είπαν οι προλαλήσαντες και η κυρία Κράτσα Μπίλτα αναφέρθηκε στο λιανικό εμπόριο. Και χαίρομαι γιατί πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό. 11% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ είναι από το λιανικό εμπόριο και 15% της απασχόλησης οφείλεται στο λιανικό εμπόριο. Δεν πρέπει λοιπόν να το αγνώμε αυτό. Στην ε, τελευταία συνάντηση της ε, Επιτροπής μας συζητήσαμε τις βέλτιστες πρακτικές και προσπαθήσαμε να δούμε τι γίνεται με ένα πρόγραμμα που έχει να κάνει με τους νέους επιχειρηματίες. Υπήρξε ένας διαγωνισμός αυτό που κέρδισε πήρε 10.000 ευρώ για να μπορέσει ακριβώς να αρχίσει μια νέα επιχείρηση. Τέτοιε πρωτοβουλίες πιστεύω ότι είναι πολύ καλές και πρέπει να τις χρησιμοποιούμε γιατί δεν είναι μόνο τα μεγάλα λόγια, είναι και τέτοια πολύ πρακτικά παραδείγματα. Η Λιθουανική λοιπόν Προεδρία σκέφτεται κάτι τέτοιο για ανταλλαγή μεταξύ των χωρών μελών όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές θα ήθελα να στο, σας το ρωτήσω αυτό. Ίσως το επόμενο εξάμεινο θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε πάνω σε αυτό, ακριβώς επειδή θα επικεντρωθούμε στο λιανικό εμπόριο. Κάτι άλλο που χάρηκα πολύ που σας άκουσα να το λέτε σχετικά με την ενιαία αγορά είναι το θέμα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Υπάρχει και το θέμα των ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών, τα ηλεκτρονικά βιβλία σε ψηφιακή μορφή. Δεν θέλουμε να μείνουμε πίσω, δεν θέλουμε αυτοί που έχουν χρήματα να μπορούν να πάρουν γνώση, να ενημερώνονται, ενώ οι άλλοι που δεν έχουν χρήματα να μην έχουν αυτή τη δυνατότητα. Γι' αυτό και οι βιβλιοθήκες θα πρέπει να είναι ένας δημόσιος χώρος στον οποίο όλοι να έχουν πρόσβαση. Να δούμε λοιπόν το θέμα του copyright τι γίνεται με όσους έχουν προβλήματα όρασης, πώς και αυτοί θα έχουν πρόσβαση σε τέτοιες βιβλιοθήκες. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να έχουν όλοι πρόσβαση στο ηλεκτρονικό βιβλίο. Και για την ψηφιακή ατζέντα, ναι, χάρηκα που σας άκουσα και εμείς προσβλέπουμε σε συνεργασία μεταξύ μας. Κύριε Πρόεδρε, πριν ο, έρθει ο κύριος Σβάμπ. Ήσασταν ο μόνος ε, άντρας μέλος της Επιτροπής ε, εδώ. Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε τις συζητήσεις αυτές και ειλικρινά λυπάμαι που δεν είναι περισσότεροι ευρωβουλευτές εδώ παρόντες γιατί είναι πολύ σημαντικό. Είμαστε στην αρχή της Λιθωνικής Προεδρίας και πρέπει να μπουν τα πράγματα σωστά. Α, βλέπω ότι φοράτε και το μπλε σας φουλάρι, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Σαλντεμόζο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τον Υπουργό που ήρθε σήμερα να συζητήσουμε. Χαίρομαι και εγώ, λοιπόν, που λέτε ότι είστε διατεθειμένος να συνεργαστείτε μαζί μας. Γιατί έχουμε πολλά θέματα μπροστά μας. Και όχι μόνο σήμερα, αλλά θα έχουμε κατά τη διάρκεια όλου του επόμενου εξαμήνου. Οπότε σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείχνετε. Εμείς λοιπόν στην Επιτροπή αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προσπαθούμε να δουλεύουμε σκληρά προκειμένου να ολοκληρώσουμε τα θέματά μας όσο γίνεται πιο γρήγορα. Να μπορούμε δηλαδή να ξεκινάμε τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, να, για παράδειγμα για την ασφάλεια των προϊόντων, όσο γίνεται πιο γρήγορα. Είναι μια πολύ βασική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί έτσι μπορούμε απτά να δείξουμε στους Ευρωπαίους πολίτες ότι η Ευρώπη μπορεί να κάνει τη διαφορά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι μια υπόθεση αυτή που μας απασχολεί όλους. Έχω λοιπόν δύο πράγματα να ρωτήσω για την ασφάλεια των προϊόντων. Μια μεγάλη συζήτηση που γίνεται εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει να κάνει με την προέλευση του προϊόντος ποια είναι η προέλευση του προϊόντος. Στο Συμβούλιο τι γίνεται με αυτό που έχει ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ένδειξη αυτή της προέλευσης του προϊόντος θα είναι τελικά υποχρεωτική ή όχι. Η ετικέτα made in θα είναι υποχρεωτική. Ξέρω ότι γίνονται ακόμα συζητήσεις, εμείς όμως πιστεύουμε ότι πρέπει να τοποθετηθείτε πάνω σε αυτό. Και υπάρχει και κάτι άλλο που έχει να κάνει με αυτά που έλεγε η κυρία Ρούλε νωρίτερα. Το θέμα των ε, πόρων που έχουμε για την εποπτεία της αγοράς είναι δύσκολο και το ξέρουμε. Είναι δύσκολο να πείσουμε το Συμβούλιο να διαθέσει αρκετά κονδύλια για να ελέγξει την αγορά. Είναι όμως αποφασιστική σημασία για μας τους Ευρωβουλευτές. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχουν αρκετοί πόροι που να προορίζονται ειδικά στον έλεγχο της αγοράς. Γιατί δεν έχει νόημα να έχουμε μια πολύ γερή νομοθεσία, αν από την άλλη μεριά δεν μπορούμε να την θέσουμε σε εφαρμογή. Τι γίνεται λοιπόν, πού βρίσκεται η συζήτηση αυτή στο Συμβούλιο. Εσείς αντιλαμβάνεστε τα επιχειρήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και θέλω να προσθέσω και κάτι ακόμα. Στη δικιά μου τη χώρα, στη Δανία, μάθαμε και δίνουμε περισσότερα κονδύλια για τον έλεγχο της αγοράς από ό,τι κατά το παρελθόν, ιδιαίτερα για τα ηλεκτρικά ε, μηχανήματα, για τα παιχνίδια, για τα πρώτα υγιεινής. Είναι ένα παράδειγμα από το οποίο μπορείτε και εσείς να εμπνευστείτε. Ξέρω βέβαια κύριε Υπουργέ ότι αυτό θα είναι αποφασιστική σημασία για το Κοινοβούλιο και που θα κάνει την υπόθεση να πάρει τον έναν ή τον άλλο δρόμο. Γιατί είναι μια πολύ βασική προϋπόθεση συνεκβάμουν προκειμένου να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία μαζί σας. Είμαστε διατεθειμένοι να προχωρήσουμε σε συμβιβασμούς, αλλά να ξέρετε ότι και εμείς έχουμε σημαντικά θέματα. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Δείξατε από την αρχή του εξαμήνου σας ότι είστε διατεθειμένος για συνεργασία και ελπίζω τα αποτελέσματα να είναι στο ύψος των προσδοκιών μας. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε κυρία Σαλουμόζε. Σίγουρα και εσείς και κύριε Πίτη Κάνεν έχετε πολύ σημαντικό ρόλο να, παίξετε σε αυτή την υπόθεση. Ο κύριος τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και με συγχωρείτε που καθυστέρησα. Κύριε Υπουργέ, χαίρομαι ιδιαίτερα που είσαστε μαζί μας σήμερα. Όλοι είμαστε, αν θέλετε, εμπλεγμένοι και στην προεκλογική εκστρατεία για τις εκλογές, τις ευρωεκλογές ε, του που υπέρχονται. Αλλά αξιολογήσετε θετικά την έκθεση για την εσωτερική αγορά και ήταν πολύ καλό αυτό, αλλά πρέπει να πούμε ότι η πλειονότητα των συναδέλφων πιστεύουν ότι θα πρέπει να κάνουμε πιο πολλά προκειμένου αυτά που αποφασίζονται στο Κοινοβούλιο να φτάνουν τελικά πιο άμεσα στους πολίτες. Και η πολιτική στάση στην Επιτροπή και η στάση ενδεχομένω και του Συμβουλίου σε κάποιες περιπτώσεις τελικά οδηγούν στο να παρεμποδίζεται και να, αν θέλετε, επιβραδύνεται ο αντίκτυπος αυτός ε, του σκληρού έργου που αποφασίζεται μετά από μεγάλες διαδικασίες σε ό,τι αφορά δηλαδή τον αντικτύπο στον πολίτη. Θεωρώ ότι θα είναι δύσκολος ο δρόμος μπροστά γιατί σε κάθε χώρα ασφαλώς θα υπάρχουν κάποιες ε, αντιρρήσεις για τις ενιαία εφαρμογή αυτών που αποφασίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επειδή Πάντα είναι πιο δημοφιλές να παρουσιάζει κανείς νέες προτάσεις παρά να εφαρμόζει σωστά ε, τα παλιά νομοθετήματα. Σας ευχαριστώ λοιπόν που θίγετε το θέμα αυτό και νομίζω ότι το Κοινοβούλιο και με τα μικρά και με τα μεγάλα κρατημέρια και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να φροντίσει προκειμένου να καταλήγουμε τελικά σε πιο καλά αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ λέει ο για τις ερωτήσεις αυτές που θέσατε και θα δώσω το λόγο στον Υπουργό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να απαντήσω στην ερώτηση της κυρίας Στήλερ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι το ελεύθερο εμπόριο επηρεάζει πραγματικά, και το λιανικό εμπόριο, συγγνώμη, επηρεάζει πάρα πολύ την ευρωπαϊκή αγορά. Αποτελεί, αν θέλετε, το, βασικό, παράγοντα που δημιουργεί θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. Έχετε απόλυτο δίκιο σε ό,τι αφορά το ΑΕΠ και το 15% των θέσεων εργασίας. 33 εκατομμύρια άνθρωποι, ξέρετε, απασχολούνται στον κλάδο αυτή. Είναι τεράστιος ο κλάδος και δυστυχώς ο αριθμός των τομέων σε ό,τι αφορά την μεταφορά υπηρεσιών και αγαθών διασυνοριακά εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλος τομέας που να παρεμποδίζει, να παρεμποδίζεται. Και έχετε δίκιο ότι εδώ υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Στις αρχές του έτους προτάθηκε ένα σχέδιο για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα του λιανεμπορίου. Και χαίρομαι που αναφέρω ότι η σημασία του θέματος αυτού τονίζεται ιδιαίτερως και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προσβλέπουμε σε όσο μεγαλύτερη συνεργασία και υποστήριξη από πλευρά σας γίνεται. Η Λουθιονική Προεδρία προγραμματίζει να συμπεριλάβει στα συμπεράσματα του Συμβουλίου κάποια εκτίμηση σε σχέση με την, το ρόλο του λιανεμπορίου. Και θα συσταθεί μια ειδική ομάδα εργασίας για να λάβει πιο συγκεκριμένα μέτρα. Ρωτήσατε επίσης σε ό,τι αφορά τις βέλτιστες πρακτικές. Όντως η ατζέντα μας περιλαμβάνει εκδηλώσεις σχετικές. Το Νοέμβριο, δεν το ανέφερα, το Νοέμβριο όμως θα συνέλθει μια ε, επιλογή, θα είναι μια εκδήλωση όπου και θα απονεμηθούν βραβεία σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τις καλύτερες ε, συνέργειες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Και στην εκδήλωση αυτή νομίζω ότι θα έχουμε μια καλή πλατφόρμα για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και βέλτιστων εμπειριών. Επίσης, μιλήσατε για τα ηλεκτρονικά βιβλία. Συμφωνώ μαζί σας ότι πρόκειται για ένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική ατζέντα στην ομιλία μου αναφέρθηκα σε θέματα προώθησης της ηλεκτρονικής ατζέντα και προτιμάζουμε δύο προτάσεις για τα ηλεκτρονικά βιβλία. Θα δούμε πώς θα αναπτυχθεί πιο ταχαίως, αν θέλετε, ο κλάδος αυτός στα πλαίσια της ηλεκτρονικής ατζέντα. Να απαντήσω τώρα στις ερωτήσεις της κυρίας Σαλτιμόζα για την ασφάλεια των προϊόντων. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε εργαστεί πάρα πολύ σκληρά σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Γνωρίζετε ποια θέματα ε, προκύπτουν από πρώτο χέρι. Σε ό,τι αφορά τώρα την τη στάση του Συμβουλίου. Να σας πω, δεν υπάρχει κάποια ενιαία στάση του Συμβουλίου. Κάποια κρατημέλη είναι υπέρ της συμπερίληψης ε, της ρήτρας αυτής στο νομοθετικό σχέδιο και κάποια άλλα κρατημέλη είναι αντίθετα. Εμείς ως Προεδρία, ως διαμεσολαβητής, αν θέλετε και μεσάζοντας, θα έχουμε ένα πολύ σημαντικό καθήκον στον, στο θέμα αυτό θα προσπαθήσουμε να το επιτελέσουμε και να βρούμε μια συμφωνία, ένα συμβασμό σε πρώτη ανάγνωση, όπως είπα και προηγουμένως. Και πριν τη λήξη της θητείας του Κοινοβουλίου. Αν όλα πάνε κατευχήν, Ελπίζουμε τον Νοέμβριο να έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία με το Κοινοβούλιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους πόρους σχετικά με την αγορά. Ένα περίπλοκο θέμα, ξέρετε. Καταρχάς, ένα θέμα του πόσα ιδρύματα, πόσα, πόσες υπηρεσίες χρειαζόμαστε σε ό,τι αφορά την αγορά και ποια θα πρέπει να είναι η κατανομή των ευθυνών τους ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος τους. Υποστηρίζουμε την άποψη ότι θα πρέπει να ενισχύθει ασφαλώς η υποπτία της αγοράς. Το δίχως άλλο. Α, ωστόσο θα πρέπει να τονίσω ότι συνεχίζεται ακόμα η σχετική συζήτηση και θα συμμετέχουμε ενεργά στη συζήτηση αυτή. Και τώρα να στραφώ στα ερωτήματα που έθεσε ο κ. Σβάπ. Σύμφωνα απόλυτα ότι τα νομοθετήματα δεν θα πρέπει να είναι κενά περιεχομένου, θα πρέπει να λειτουργούν. Να είναι εργαλεία που να λειτουργούν πραγματικά. Στην ατζέντα που σας παρουσίασα, Υπάρχει ένα light motive, αν θέλετε, ε, σε ό,τι αφορά την ανάλυση, τα συμπεράσματα και τις συστάσεις. Θα επικεντρωθούμε στο πώς εφαρμόζονται τέτοια σημαντικά νομοθετήματα. Μιλώ για την, ε, το Small Business Act και άλλες οδηγίες και θα κάνουμε και συγκεκριμένες συστάσεις για την καλύτερη εφαρμογή τους. Και τώρα θα ήθελα να στραφώ στο Συμβούλιο Ταγωνιστικότητας του Νοεμβρίου και στην διακυβέρνηση ενιαίας αγοράς και τις σχετικές πτυχές. Για το νέο Solvit, για το IMI και για τις, ε, τα single point contacts και τις σχετικές δραστηριότητε θα κάνουμε σχετικές συστάσεις. Επίσης, ρωτήσατε κατά πόσον χρειάζονται όντω νέες προτάσεις, νέα νομοθετήματα, όταν υπάρχουν διαθέσιμα νομοθετήματα τα οποία δεν εφαρμόζονται απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Καταρχά, θα πρέπει και να επικεντρώσουμε την προσοχή μα στη σωστή εφαρμογή των ήδη υφισταμένων νομοθετημάτων και μόνο σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι αποτύχουν ή δεν μπορούν να εφαρμοστούν σωστά. Τότε μόνο θα πρέπει να αναλογιστούμε την πρόταση Good. Well, um, Ευχαριστούμε πολύ που καλύψατε τόσα πολλά θέματα. Νομίζω ότι αναφερθήκατε σε όλες τις εκθέσεις πρωτοβουλίας μας. Και ένα από τα πράγματα που σίγουρα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι να έχουμε ένα συνεχή διάλογο μαζί σας φτάνουμε στο τέλος του νομοθετικού προγράμματος της θητείας μας. Πρόσφατα είχαμε μια πολύ επιτυχή επίσκεψη στη Λιθουανία και μιλήσαμε με την πρόεδρο. Ξέρω ότι σας ενδιαφέρει πάρα πολύ το να προχωρήσουμε και στο Συμβούλιο. Η Επιτροπή μας πάντως να ξέρετε ότι θα χρησιμοποιήσει ό,τι μέσα έχει στην ε, διάθεσή της, μελέτες, η έκθεση του κύριου ΣΒΑΠ για παράδειγμα, για την προστιθέμενη αξία της ενιαίας αγοράς και η Κομισιόν ετοιμάζει μια αντίστοιχη μελέτη. Όλα αυτά σίγουρα θα τα συζητήσετε κι εσείς στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας. Ελπίζω να έχουμε και άλλη ευκαιρία να έχουμε διάλογο μαζί σας. Αν μας δοθεί ευκαιρία θα τη χρησιμοποιήσουμε. Το σχέδιο αυτό του διαγωνισμού που λέτε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σίγουρα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και για μας. Για την ψηφιακή εσωτερική αγορά νομίζω το Νοέμβριο θα υπάρξει κάτι και θα συμμετέχουμε κι εμείς. Χαίρομαι που ήρθατε σήμερα, που είναι, είσαστε στην αρχή της Προεδρίας σας και ελπίζω να σας ξαναδούμε προς τα τέλη της Προεδρίας σας για να μας πείτε τι έχει γίνει όλο αυτό το εξάμεινο. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, για όλες τις απαντήσεις σας. Ένα θερμό χειροκρότημα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Η σημερινή συνάντηση που είχα μαζί σας πρέπει να ξέρετε ότι ήταν για μένα μια πολύ σημαντική ευκαιρία. Ήταν πολύ χρήσιμο που άκουσα τις δικές σας απόψεις και τις δικές σας προτάσεις. Και πιο σημαντικό ακόμα, άκουσα ότι με στηρίζετε και υποσχεθήκατε να συνεργαστούμε. Αυτό για μένα έχει μεγάλη σημασία. Ε, να ξέρετε ότι και εμείς από τη Λιθουανική Προεδρία προσβλέπουμε σε καρποφόρα συνεργασία μαζί σας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ωραία, κλείνουμε αυτό το σημείο. Θα αποχαιρετήσω τον Υπουργό και θα συνεχίσουμε 4,5 με τα επόμενα θέματα. Είναι δικιά μου έκθεση, οπότε ναι, θα γυρίσω, μην φοβάστε. Θα είμαι πίσω στις 4.30 για να έχω και ένα καλό ακροατήριο. So, ladies and gentlemen, can we now move on to the next item? Is that okay? Να περάσουμε στο επόμενο θέμα, συνάδελφοι. Παρακαλώ, καθίστε. Uh, um, Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, να προχωρήσουμε και να περάσουμε στο σχέδιο γνωμοδότησής μου για την Επιτροπή Βιομηχανίας, αν συμφωνείτε. Και είναι λίγο ασυνήθιστο ως διαδικασία, αλλά θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι οι συνάδελφοι στην Επιτροπή Βιομηχανίας ήταν πάρα πολύ πρόθυμη. ήθελα να κάνω μια τέτοια έκθεση εφαρμογής για τις ηλεκτρικές, επικοινωνίε. επικοινωνίες. είναι πάρα πολύ ενθουσιώδη για το θέμα αυτό. Το θέμα αυτό ξέρετε θα περιλαμβάνει διάφορες ε, συνδεδεόμενε οδηγίε, οι οποίες όλες συνδέονται σε ένα πακέτο και εντάσσονται σε ένα σε μια οδηγία πλαίσια για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τις τηλεπικοινωνικέ και σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα του καταναλωτή. Και αυτά, ξέρετε, ήταν πάντα δική μας ε, αρμοδιότητα. Είχα λοιπόν ε, την τιμή να είμαι εισηγητή για την πρώτη αναθεώρηση του πακέτου αυτού το 2002, ε, δεν κάνω λάθος, και για την επόμενη αναθεώρηση που συμφωνήθηκε το 2009. Και φυσικά ήμουν, με ενδιέφερε ιδιαίτερα η Επιτροπή μας να συμμετέχει και να συμβάλλει στην έκθεση της κυρίας Στράτμαν. Γιατί θα ακούσατε ότι όταν ήρθε να μας μιλήσει η κυρία Κρούς πριν από κανένα μήνα, μας παρουσίασε ένα πάρα πολύ φιλόδοξο σχέδιο σε ό,τι αφορά πολιτικές πρωτοβουλίες πριν τη λήξη της θητείας και σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα θέματα προαγωγής και άλλα θέματα προστασίας του καταναλωτή και σε ό,τι αφορά την ιδιωτερότητα των δικτύων. Νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά αφορούν ιδιαίτερα την Επιτροπή Βιομηχανίας αλλά και εμάς. Γι' αυτό λοιπόν συμφωνήσαμε σε μια τέτοια πιο συνοπτική διαδικασία και λυπάμαι ιδιαίτερα που η γνωμοδότηση δεν πρόφασε να μεταφραστεί, ήταν στα αγγλικά μόνο, αλλά θεωρώ ότι ήταν πιο καλό να γίνει αυτό παρά να μην υπάρξει καμία γνωμοδότηση. Και επίση είναι πάρα πολύ σημαντικό η Επιτροπή μα με το ιστορικό μα σε ό,τι αφορά την υποστήριξη προστασία των καταναλωτών. Ιδιαίτερω επειδή υπάρχουν και πάρα πολλέ τέτοιε πρωτοβουλίε στο πακέτο που συμφωνήθηκε το 2009 για τι καταναλωτικές υπηρεσίε, ήταν σημαντικό λοιπόν να δοθεί και η δική μας ε, η άποψη. Τι αποφασίσαμε λοιπόν να κάνουμε μαζί με τους κοιόντες εισήγητης ε, παρά να βιαστούμε και να κάνουμε μια ψηφοφορία τώρα, αυτή την εβδομάδα, να κάνουμε και να καταβάλουμε, να υποβάλουμε τροπολογίες τέλη Αυγούστου και να ψηφίσουμε το Σεπτέμβριο η Επιτροπή Βιομηχανίας θα ψηφίσει, αν δεν κάνω λάθος, τέλη Σεπτεμβρίου. Ναι, σωστά. Ναι, 25 και 26 Σεπτεμβρίου. Και πρόφανως ε, θέλουμε να μας ανακοινώσει η Επιτροπή Κρούς ε, ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει. Γι' αυτό λοιπόν κάναμε αυτά και ακολουθήσαμε αυτή την, ε, αν θέλετε, περικεκομένη διαδικασία. Έχετε λοιπόν το αγγλικό κείμενο μπροστά σας. Ήμουν σαφέστατος εδώ. Νομίζω ότι καλύπτω μόνο τις πτυχές επί των οποίων είχε συμφωνήσει η αρχική πρόταση της Επιτροπής μας. Και έχω την αίσθηση ότι σε διάφορα θέματα, σε διάφορα τον καταναλωτή, θα πρέπει να δώσουμε μια όθεση στις ε, ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών, προκειμένου με ενιαίο τρόπο να εφαρμόσουν τις ρήτρε για την προστασία του καταναλωτή. Ξέρω ότι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες σε κάποια κρατημέλη, γιατί κάποια κρατημέλη και τα σχετικά υπουργεία για την προστασία του καταναλωτή συμμετέχουν πιο έντονα και σε κάποιες περιπτώσεις, ξέρετε, αυτό αποδυναμώνει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να το δούμε αυτό στα πλαίσια του κανονισμού για, την ηλεκτρονική, τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. προσέθεσα επίσης κάποια θέματα για κάποιες τάσεις που διαγράφονται στην αγορά. Κάποιες τάσεις μετά το 2009 είναι, ξέρετε, ένας ταχαίως μεταβαλλόμενος τομέας και θεωρώ ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες αυτές οι μεταβολές στις ε, ρυθμίσεις για την προστασία των καταναλωτών. Νομίζω ότι ξέρετε Ξέρετε, αυτά τα συμβόλαια που υπάρχουν, τα οποία δεν αποτελούν συμβόλαια δέσμες. Μιλάμε επίσης για θέματα παροχής υπηρεσιών και θέματα όπως το, η διάρκεια ισχύω του της σύμβασης, μία σαφής ενημέρωση για το τι περιλαμβάνεται ή όχι και ενημέρωση του καναλωτή για τη διάρκεια ισχύω και την καταγγελία μιας σύμβασης, ε, θέματα επιδοτήσεων, πρόορες καταγγελίας ε, σύμβασης ε, τι γίνεται όταν καταγγέλει, πούμε, όταν διακόπτει κανείς μια σύμβαση πρόωρα, αλλά έχει πάρει ένα τηλέφωνο, έναν υπολογιστή στα πλαίσια της σύμβασης. Η μη διακριτική μεταχείριση. Όλα αυτά λοιπόν καλύπτονται και ιδιαίτερως στο γενικότερο πλαίσιο της διαφάνειας της σύμβασης, όπως την αποκαλώ. Υπογραμμίζω επίσης επίσης την δυνατότητα που πρέπει να έχει ο καταναλωτής να αλλάξει πάροχο, γιατί θεωρώ ότι αυτό αποτελεί βασικό στοιχείο μιας δυναμικής αγοράς και στην, στο θέμα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Το γεγονός ότι μπορεί κανείς να μεταφέρει τον αριθμό του, για παράδειγμα, σε ένα άλλο πάροχο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στην ε, αναθεώρηση του 2009, το Κοινοβούλιο ζήτησε κατεπηγόντως μεγαλύτερη κινητικότητα. Και κάπως νομίζω απογοητευτήκαμε από την έκθεση που λάβαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φαίνεται ότι δεν είναι όλες οι χώρες σε θέση να πούν ότι πληρούν όλους τους στόχους αυτούς κινητικότητας. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να εφαρμοστούν. Επίσης, φορητότητα, συγγνώμη. Μιλάμε επίσης ε, για την ίση πρόσβαση σε χρήστες με αναπηρία. Νομίζω ότι και πάλι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Υπάρχει μια συγκεκριμένη πτυχή σε ό,τι αφορά τον εβραίος διαδεδομένο αλλά και αν θέλετε πολύ παρεξηγημένο όρο της ουδετερότητας δικτύου. Εμείς αποφεύγουμε αποφύγαμε να χρησιμοποιήσουμε στην οδηγία του 2009 τον όρο αυτό, γιατί ειλικρινά κανείς δεν μπορούσε να συμφωνήσει τι ακριβώς σήμαινε. Και θεωρούμε ότι αυτό εξακολουθεί να ισχύει. Κάποιοι μιλούν για ουδετερότητα δικτύου και εννοούν ότι οι πάροχοι δεν επιτρέπουν να παρέχονται ε, υπηρεσίες όπως το IPE, voiceover, ε, το Skype για παράδειγμα. Αυτό όμως δεν είναι η ουδετερότητα δικτύου. Αυτό έχει να κάνει με μια συμπεριφορά η οποία είναι αντιανταγωνιστική αν θέλετε. Το θέμα με την ουδετερότητα δικτύου έχει να κάνει με το γεγονός ότι η ποιότητα των υπηρεσιών και των αγαθών ενδεχομένως να σημαίνουν ότι ο πάροχος κάνει μια διακριτική μεταχείριση προς κάποιους καταναλωτές που χρησιμοποιούν τα δικά τους προϊόντα. Και αυτό λοιπόν μας απασχολεί ιδιαίτερως και δώσαμε στους νομοθέτες σαφή εργαλεία για να μπορούν να παρέμβουν σε περίπτωση που διαπιστώνουν ότι υπάρχει τέτοια διακριτική μεταχείριση. Και επίσης σε συνδυασμό με συμβάσεις πιο διαφανείς εξ αρχής θεωρούσαμε ότι έχουμε δώσει πολύ σημαντικά εργαλεία στους νομοθέτες και οι νομοθέτες όντω δηλώνουν ότι έχουν τα εργαλεία αυτά πλέον στα χέρια τους, αλλά δεν είμαστε σίγουροι κατά πόσον τα χρησιμοποιούν επαρκώς. Δεν είναι καλό λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει οποιαδήποτε άλλη πρόταση, γιατί καταδεικνύεται ότι τα εργαλεία που υπάρχουν σήμερα είναι αρκετά ικανοποιητικά. Το θέμα είναι κατά πόσον εφαρμόζονται επαρκώς. Ίσως να χρειάζονται μεγαλύτερη παρότρινση οι νομοθέτες για να τα χρησιμοποιήσουν πιο αποτελεσματικά. Πολλοί από εσά ήσασταν εδώ την προηγούμενη Πέμπτη. Έγινε μια πολύ καλή συζήτηση για το ψήφισμα για την ψηφιακή ενιαία αγορά και για την χρήση του αριθμού 112 πανευρωπαϊκά. Κοιτάξτε, υπάρχουν ακόμα κάποιες χώρες που δεν έχουν εφαρμόσει όλες τις διατάξεις. Και τέτοια στοιχεία που είχαν συμπεριληφθεί ήδη το 2002. Και η Επιτροπή μας είχε θέσει το ερώτημα για τους αριθμούς 116 για κοινωνικές υπηρεσίες ουσιαστικά, για γραμμές εξυπηρέτησης του πολίτη, ενημέρωσης του πολίτη, Υπάρχει και μια ιδιαίτερη γραμμή για τα αγνοούμενα παιδιά 116.000. Θεωρώ ότι αυτά δεν έχουν ακόμα εφαρμοστεί επαρκώ σε όλε τι χώρε. Κάτι άλλο κάνω να σας αναφέρω, γιατί πολύ εξήμων θα θυμάστε ότι κάναμε μία συζήτηση για έναν χώρο για ευρωπαϊκά, για ευρωπαϊκά τηλέφωνα, για Ευρωπαϊκού τηλεφωνικού αριθμού. και κάποιους αριθμούς 3, 8, 8, 3 που θα ίσχυαν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν έχουν ακόμα χρησιμοποιηθεί αυτές οι δυνατότητες και εμείς είχαμε πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε περίπτωση που δεν έκανε τίποτα η ίδια, ίσως θα έπρεπε να φροντίσει να τα αναθέσει σε κάποιου ιδιωτικού φορεί σε κάποιες ιδιωτικέ επιχειρήσεις. Αλλά φαίνεται ότι πρέπει να υπάρχει ακόμα έλλειψη ζήτηση. Περιορίστηκα λοιπόν σε έκταση γιατί ήταν γνωμοδότηση, αλλά ελπίζω να έχω και συμμετοχή από τις ε, άλλες πολιτικές ομάδες. Μέχρι τώρα η κυρία Οχέιν νομίζω ότι είναι η μοναδική ε, στη Σιγήτρια. Δεν είμαι βεβαίως κατά πόσο οι σοσιοδημοκράτες σκοπεύουν να ορίσουν κάποιον ως σκιώτη ή εισηγήτρια. Δεν είμαι βεβαιως κατά πόσον οι σοσιαλδημοκράτες σκοπεύουν να ορίσουν κάποιον ως σκιώδη εισηγητή. Αλλά ασφαλώς όποιος θέλει να καταθέσει τροπολογίες μπορεί να το πράξει. Αυτά λοιπόν ενημερωτικά. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στην κυρία Φερχέγεν και οποιοδήποτε άλλος συνάδελφο θέλει να πάρει το λόγο ευχαρίστω να τον λάβει. Βλέπω ότι έχουμε και μια ισχυρή αντιπροσωπή από τη Γενική Διεύθυνση Connect. Θα λάβουν και αυτή το λόγο. Αλλά πρώτα η κυρία Φερχέιεν και οποιοδήποτε άλλο επιθυμεί στη συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Φερχέιεν. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Η συνεργασία μαζί σας ως εισηγητή ήταν πραγματικά πάρα πολύ ικανοποιητική και γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω. Στην έκθεση αναφέρονται πολλά και σημαντικά στοιχεία. Και σε ό,τι αφορά τις μεμονωμένες περιγραφές, εξηγείται τι σημαίνει για παράδειγμα η ουδετερότητα δικτύου, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει στο σημείο αυτό να διευκρινίσουμε ότι σε ό,τι αφορά το traffic management υπάρχουν και πάρα πολλά εμπόδια στον ανταγωνισμό τα οποία μπορούν να εγερθούν και πρέπει να εξετάζουμε τι συνέβαινε ως τώρα σε ό,τι αφορά την διακίνηση δεδομένων και επίσης ε, στα πλαίσια των best efforts ότι η καλύτερη δυνατή προσπάθεια δηλαδή με τους ε, υπάρχοντες όρους. Θα πρέπει να φροντίσουμε στα νέα επιχειρηματικά μοντέλα να μην προκύψει bundling αυτό το αναφέρεται με σαφήνεια στην έκθεση, γιατί έτσι θα δημιουργηθεί συγκέντρωση στην αγορά, συγκέντρωση περιεχομένου και στράφλωση του ανταγωνισμού. Νομίζω ότι θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι αφενός μεν υπάρχει δικτύου υπάρχουν, αλλά και δραστηριοποιούνται στον αγορά του περιεχομένου αλλά δεν θα πρέπει ποτέ να προκαλούνται στρεβλώσεις. Ένα θέμα το οποίο θα ήθελα να προσθέσω και το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην έκθεση είναι τα personal hotspots και οι σχετικές δυνατότητες, τα οποία συχνά μπλοκάρουν οι εταιρείε. Δηλαδή, παρά το γεγονό ότι έχω μια σύμβαση ανταλλαγή δεδομένων ω άτομο, ω ιδιώτη, δεν μπορώ να συνδεθώ με ένα hotspot. Καταπιέζεται, αν θέλετε. Ε, μάλλον ε, κλείνει η πρόσβαση προκειμένου να καταναγκαστεί ο καταναλωτής να κάνει και άλλη σύμβαση. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε στην έκθεση για την εφαρμογή του πακέτου τηλεεπικοινωνιών να δούμε ποιες είναι οι τεχνολογικές δυνατότητες που έχουμε ή πλέον πρόσφατες μετά την εφαρμογή της οδηγίας, ποιες ενδεχομένως προσθήκες να πρέπει να γίνουν προκειμένου και στο μέλλον να έχουμε σωστές προτάσεις οι οποίες θα προσαρμόζονται στις σημαντικές τεχνολογίες για να μην περιορίζεται η παροχή υπηρεσιών και να μην προκαλείται αδιαφάνεια για τον καταναλωτή. Το θέμα των συμβάσεων είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον καταναλωτή. Σε πολλές περιπτώσεις η ουδετρότητα δικτύου έχει να κάνει με το κατά πόσον υπάρχει διαφάνεια σύμβαση ή όχι. Τι προσφέρει πραγματικά μια σύμβαση στον καταναλωτή. Και για παράδειγμα, η αναφορά του όγκου ανά δευτερόλεπτο δεν είναι απαραίτητα ε, αξιόπιστη βάση για την σύναψη μιας σύμβασης. Νομίζω ότι στο πακέτο τηλεπικοινωνιών θα πρέπει να σκεφτούμε σε ένα άλλο κομμάτι, αν θέλετε, στην ε, οδηγία για τις καθολικές υπηρεσίες θα πρέπει να κάτσουμε να κοιτάξουμε κατά πόσον ευκρινίζεται ότι οι υπηρεσίε τηλεπικοινωνιών στον κινητό τομέα μπορούν να συμπεριληφθούν ως αναπόσπαστο κομμάτι της οδηγίας ε, καθολικών υπηρεσιών. Πρέπει να υπάρχει μια βασική πρόσβαση στο ευρυζωνικό φάσμα. Νομίζω ότι οι συνάδελφοι ενδεχομένως τις επόμενες εβδομάδες θα κάνουν παρατηρήσεις αναμφίβολα και ίσως θα μπορούσαμε να τις ε, ομαδοποιήσουμε και να σας τις υποβάλουμε εξ ονόματος του, της ομάδας του ΕΛΚ προκειμένου και μετά τις θερμινές διακοπές να μπορέσουν να συμπεριληφθούν στο σχέδιο γνωμοδότησης και να μπορέσουμε να την ολοκληρώσουμε επιτυχώς. Ευχαριστώ. Good. Well, thank you very much. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις παρατηρήσεις. Ξέρω ότι έχετε δουλέψει κι εσείς αρκετά για το θέμα αυτό, γιατί μαζί δουλέψαμε. Είναι ένα τομέα πολιτικής που μας ενδιαφέρει πολύ και ελπίζω να επιτελέσουμε πρόοδο. Κάποιος άλλος από τις πολιτικές ομάδες της υπόλοιπες θέλει να πει κάτι για την σημερινή μας συζήτηση. Ιδάλλως να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποιος θέλει να παρέμβει. Από την DG Connect. Ωραία, μπορείτε να συστηθείτε. Ευχαριστώ. Από την ε, Γενική Διεύθυνση Connect. Ευχαριστώ για την ευκαιρία να σας αναφέρω τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το σχέδιο γνωμοδότησης, για την οδηγία πλαίσιο και τις τηλεπικοινωνίες. Λίγα μόνο σχόλια για όσα είπατε για τη συνολική αναθεώρηση του πλαισίου. Όπως είπατε, τα κράτη -μέλη στα κράτη-μέλη προτάθηκε το, η μέτρων για το 2013 και υπάρχουν κάποια πρώτα συμπεράσματα και κάποια ζητήματα στα οποία χρειάζεται καταπήγουσα δράση. Είναι πολύ δύσκολο ακόμη να οργανώσουμε σφαιρική αναθεώρηση σε αυτή τη φάση, γιατί μόλι το 2009 εγκρίθηκε, αλλά στο πλαίσιο της προετοιμασίας της επόμενης θητεία της Ευρωπαϊκή Επιτροπής θα ε, φροντίσουμε να υπάρξει μια σφαιρική εξέταση του πλαισίου. Θα χρειαστεί να περάσουν χρόνια για να γίνει η θεώρηση και να ολοκληρωθεί, αλλά κάποια ζητήματα χρειάζονται κατεπίγουσα προσοχή. το τεράστιο δυναμικό της ψηφιακής οικονομίας ως ε, πηγή ε, καινοτομία, ε, δημιουργία θέσεων απασχόληση και οικονομική ανάπτυξη, ακόμη δεν έχει εξοπλιστεί πλήρω γιατί δεν έχουμε μια ενιαία αγορά για τη τηλεπικοινωνίε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω είδαμε τι γίνεται με την προοπτική ολοκληρωμένη αγορά για τι τηλεπικοινωνίε, θα μπορούσαμε να έχουμε 110 δι ευρώ κέρδο ετησίω. Και σκοπεύουμε, όπω σημειώνεται και στα συμπεράσματα του Ερενού Συμβουλίου, να προτείνουμε συγκεκριμένα μέτρα για να αρθούν οι φραγμοί για τέτοια ενιαία αγορά. Η ενιαία αγορά για τι τηλεπικοινωνίε σημαίνει επί τη ουσία να επιτρέψουμε στου πολίτε και τι επιχειρήσει να απολαύσουν πλήρω τι τηλεπικοινωνιακέ και ψηφιακέ υπηρεσίε οπουδήποτε και αν βρίσκονται στην Ευρώπη. Να επιτρέψουμε στου παρέχοντε να προσφέρουν ψηφιακέ υπηρεσίε σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ολόκληρη την επικράτειά τη όπου και αν είναι καταχωρημένη, και να τονώσουμε βεβαίως την, την οικονομία ευρύτερα, ώστε να υπάρχει ε, μεγαλύτερη επιλογή, στην επιλογή, μεγαλύτερη επιλογή μεταξύ των ψηφιακών υπηρεσιών σε ένα όλο ένα περισσότερο ηλεκτρονικό περιβάλλον και σε ό,τι αφορά τι ιδιωτικέ παροχέ αλλά και τι ε, κρατικέ υπηρεσίες. Συμφωνούμε μαζί σα ότι οι καταναλωτές θα, θα πρέπει να βρισκόνται στο κέντρο των ε, μέτρων που προτείνουμε λόγου χάρη, όπως και ο Αντιπρόεδρος η Αντιπρόεδρος Κρούς ε, επεσήμανε σε ομιλία της αυτή την Επιτροπή πρόσφατα, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τα τέλη της περιαγωγή. Και θα συμφωνήσω με τον κύριο Χάρμπορ ότι ένα συνεκτικό πλαίσιο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαραίτητο προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια και να μπορεί κανείς να αλλάξει παροχέα. Έτσι θα φροντίσουμε αυτά να βρίσκονται στην καρδιά τη πρότασή μα. Θα ολοκληρώσω ευχαριστώντα σα για την πρόθεσή σα να στηρίξετε τον Αντιπρόεδρο Κρού, η οποία ενθαρρύνεται ιδιαίτερω από τι τάσει σα. Ε, Στι επερχόμενε συνομιλίε για την πρωτοβουλία αυτή. Ευχαριστώ. Well, thank you for that contribution. Σας ευχαριστώ. Από την άποψη της ανθεώρησης, να πω ότι η πρώτη ρήτρα που έχω, το πρώτο εδάφιο της νομοδότησης, σε συνδυσμό με όσα η κυρία Τροτμάν κάνει στην Επιτροπή Βιομηχανίας, αναφέρεται ακριβώς αυτό. Δεν ήταν το θέμα να το αναφέρουμε ξεχωριστά εδώ, απλώς να δείξουμε ότι συμβαδίζουν οι απόψεις μας καθώς θέλουμε ακριβώς μια τέτοια αναθεώρηση για το πλαίσιο που είχε δημιουργηθεί για το 2007-2013 και υπάρχει και ένα επιπλέον εδάφιο που αφορά το ευρωζωνικό, τις ευρωζωνικές υπηρεσίες κάτι που συμπεριλαμβανόταν μεταξύ των προτασεών μου και που είχατε την ευκαιρία να το δείτε. Ναι, είναι και ενδιαφέρον αλλά και διασυνδέει τη δική μας δουλειά για την παροχή οικουμενικών υπηρεσιών και τις ε, επενδύσεις καθώς και την πρόσβαση σε υποδομές που αναφέρονται και στην έκθεση της κυρίας Τροτμάν. So... Ναι. Σας διαβεβαιώ ότι όλα αυτά θα οδεύουν παραλληλώς. 28 Αυγούστου ε, η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών και αν άλλε πολιτικέ ομάδε θέλουν να συνεισφέρουν, ευχαρίστω. Θα το συζητήσουμε και θα ψηφίσουμε στι 5 Σεπτεμβρίου. Ωραία. Θα προσπαθήσω να συγκαλέσω συνάντηση για όλους όσοι ενδιαφέρονται αφού επιστρέψουμε μετά τις θερινέ διακοπέ. Right. Ωραία. Ας προχωρήσουμε. Επόμενο θέμα. Και αυτό έχει να κάνει με την ενιαία ψηφιακή αγορά. Ηλεκτρονική ταυτοποίηση και υπηρεσίε εμπιστοσύνη. Για ηλεκτρονικέ συναλλαγέ στην εσωτερική αγορά. Η συγκέντριά μα είναι η κυρία Γκαλό γνωμοδότηση της Επιτροπής ε, Βιομηχανίας πρέπει να εγκριθεί αύριο, διότι η Επιτροπή Βιομηχανίας θα ψηφίσει τη δική της έκθεση στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου και θα πρέπει να δούμε και τις συμβαστικές τροπολογίες που έχουν ετοιμαστεί. Νομίζω όλοι θα πρέπει να τις έχετε λάβει. Είναι περίπου 14 νομίζω. Για να δούμε ποιοι είναι εδώ από τους κοιόντους εισηγητές, η κυρία Πέντεργαστ. Από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες υπάρχει κάποιος εκ μέρους της. Ο κύριος Μπουζόη έφυγε, ο κύριος Κρόιτσμαν θα αναλάβει, ο κύριος Έμστρομ δεν είναι εδώ. Είμαι εγώ εδώ όμως, οπότε μεταξύ μας θα τα βρούμε. Και θα μπορέσει να απαντήσει κάποιος στην κυρία Γκαλό. Παρακαλώ αυτό το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ξεκινήσω ευχαριστώντας όλους τους αδελφούς που μου έδωσαν τα φώτα τους και τη στήριξή τους. Μου ξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τις συμβαστικές τροπολογίες που έχουμε συντάξει από κοινού. Θα αναφερθώ στα σημεία όπου υπήρξε συμφωνία, αλλά δεν θα τα εξαντλήσω. Πρώτο σημείο, Εργαστήκαμε πολύ για να επαναδιατυπωθεί το άρθρο 2, εδάφιο 1 και 2, που αφορά το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Όντως, χρειαζόταν μια σαφής νομική βάση που να διασκεδάζει τις νομικές αβεβαιότητες της αρχικής εκδοχής του κειμένου, όπως το είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλαμε να καθορίσουμε τους όρους της αμοιβαίας αναγνώρισης ώστε να είναι αποτελεσματική. Μιλάμε πάντα για ηλεκτρονικά συστήματα ταυτοποίησης που έχουν κοινοποιήσει και θεσπίσει τα κράτη-μέλη και για τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης, τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες εμπιστοσύνης. Το δεύτερο σημείο στο οποίο καταλήξαμε σε συμφωνία έχει να κάνει με την ε, συμπερίληψη δύο νέων άνθρων ένα πρώτο άρθρο που είναι ουσιαστικά οδηγίες χρήσης, οδηγίες χρήσης που θα πρέπει να ακολουθούν τα κράτη-μέλη σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο κενό, κάποιο σφάλμα στο σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης ως προς την κοινοποίηση ή ως προς την ταυτοποίηση αυτή καθεαυτή. Υπάρχει κι άλλο ένα άρθρο το οποίο διευκρινίζει την ευθύνη των κρατών μελών πάντοτε ως προς τα συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Τώρα για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση να κλείσω, θυμίζοντας και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι δεν ήθελα να θέσω ένα αμφιβόλο την διαλογικότητα των συστημάτων, τη διαλειτουργικότητα μάλλον, με μέγιστες απαιτήσει ε, ασφαλεία, προκειμένου να μην ε, πληγεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής ε, ψηφιακής αγοράς. Του αντίον θεωρώ ότι με ε, τις ελάχιστες απαιτήσει ασφάλειας διασφαλίζουμε ακριβώς τη διαλειτουργικότητα. Και μάλιστα, εάν υπάρξει εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών. Έτσι θα πετύχουμε το στόχο μας και θα πάρουμε τα τελευταία εμπόδια που δεν επιτρέπουν στην ενιαία ηλεκτρονική αγορά να δημιουργηθεί. Δεύτερο τμήμα, ε, υπηρεσίες εμπιστοσύνης, ηλεκτρονικές υπηρεσίες εμπιστοσύνης. Και εδώ συνεργαστήκαμε με του συναδέλφου για να ενισχύσουμε τις νομικέ αρχές που διέπουν το κείμενο σε ό,τι αφορά την ευθύνη των ε, παρεχόντων υπηρεσίες εμπιστοσύνη στην Ευρώπη και όσων προέρχονται από τρίτες χώρες. Για αυτό το σκοπό εξετάσαμε τι έχει ήδη πάει καλά με την προηγούμενη οδηγία του 99 και επιζητήσαμε να αποσαφηνίσουμε την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τελευταία παρατήρηση, τελευταίο σημείο μάλλον, Απλούστευση. Απλούστευση για το άρθρο 17. Άρθρο που αφορά τις ενισχυμένες υπηρεσίες ή χαρακτηρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνη, καθώς και τις απαιτήσει που πρέπει να ισχύουν για αυτούς που παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες, ώστε να διευκολύνουμε το έργο των φορέων ελέγχου. Όπως το είπατε και εσείς, Πρόεδρε, 14 συμβαστικές τροπολογίες έχουμε μπροστά μας, Νομίζω ότι υπάρχει ευρεία συνένεση. Θα δούμε βέβαια τι θα γίνει αύριο. Και παραμένω στη διάθεση των συναδέλφων για να συζητήσουμε, συνομιλήσουμε, για να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση μπορεί να ανακύψει. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Uh, right. Ωραία. Ποιο θέλει να απαντήσει εκ μέρου των πολιτικών ομάδων. Κύριε Κρόιτσμαν, νομίζω έχετε πάρει το θέμα, έχετε αναλάβει εκ μέρου του κυρίου Μπουζόη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επειδή είναι ε, ευρεία η υποστήριξη όλων των μερών τη Επιτροπή, θεωρώ ότι θα μπορέσω να είμαι πολύ σύντομο. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή η λύση στην οποία καταλήξαμε. Θα έχουμε να μιλήσουμε για την πρόσβαση με ηλεκτρονικά μέτρα ταυτοποίησης. Και ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ικανοποιημένη με, την, το συμβιβασμό, με τη συμβαστική μας πρόταση, γιατί ε, αποτυπώνει και τη δική της θέση εν μέρη τουλάχιστον. Θα πρέπει να κοιτάξουμε αφενός την ε, ενιαία αγορά, αλλά και την ασφάλεια των υπηρεσιών. Δεν είναι δυνατόν με ένα διαβατήριο με ηλεκτρονική πρόσβαση, να έχουμε πρόσβαση σε ένα άλλο κράτος μέλος όπου χρησιμοποιούνται πολύ πιο πολλά τέτοια ηλεκτρονικά μέσα. Είναι επίσης σημαντικό κάποιες τεχνικές προδιαγραφές να είναι διασυνοριακές, γιατί εφόσον δεν είναι τουλάχιστον δυσανάλογες ε, στην εφαρμογή τους σε ό,τι αφορά την ευθύνη των κρατών μελών και σε ό,τι αφορά, αφορά περιπτώσεις ε, ευθύνης είναι Διαφέρει λίγο η απόψή μα σε σχέση με τι πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρώ ότι έχουμε βελτιώσει κάποια στοιχεία για καλύτερη εφαρμογή και είναι σαφέ ότι μπορούν να υποβληθούν τέτοιε αξιώσει και από ιδιώτε, εκτό και αν έχει προβλεφθεί κάτι διαφορετικό. Και σε ό,τι αφορά του παρόχου, ε, έχουμε ζητήσει μεγαλύτερη πιστοποίηση για να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια. Ελπίζω και στην Επιτροπή Βιομηχανίας όπου συνεργάζομαι επί της πρότασης αυτής να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποιες συμβαστικές προτάσεις. Δεν υπάρχει λόγος να επανεφεύρουμε τον τροχό. Σας ευχαριστώ λοιπόν συνάδελφοι και τον εισηγητή και ελπίζω οι προτάσεις μας να έχουν να σας βρουν σύμφωνους και να τις υποστηρίξετε. Ευχαριστώ. Μάλιστα λέει ο Πρόεδρος. Ως ε, σκιώδης εισηγητής ε, για την ομάδα μου, να πω ότι είναι όντω εξαιρετικέ οι συμβαστικέ τροπολογίε και ευχαριστώ πολύ την κυρία Γκαλό για την ε, προσπάθεια και τη δουλειά που έχει κάνει. Θα τη στηρίξουμε. Γιατί συνολικά η γνωμοδότηση θα είναι σημαντικότατη. Για να έχουμε ένα εύλογο και καλό αποτέλεσμα για όλο αυτό το πακέτο. Υπάρχει συμφωνία ενισχυμένη συνεργασία με την Επιτροπή Βιομηχανία. Οπότε θα περάσουν όλα αυτά απευθεία στην Ολομέλεια, χωρί ε, τροπολογία από την Επιτροπή Βιομηχανία, πράγμα που ήταν μέρο τη συμφωνία μα μαζί του. Για κάποιε πιο συγκεκριμένε πτυχέ, χαίρομαι που η κυρία Γκαλό έχει ε, προτείνει ένα σήμα εμπιστοσύνη για τι συγκεκριμένε υπηρεσίε και νομίζω ότι θα έχετε στήριξη γι' αυτό, τουλάχιστον από εμά, αλλά και από άλλους πολλούς, ε, στον κατάλογο των ψηφοριών. Επίσης για τις τροπολογίες του κυρίου Κρότσμαν για τον ιστότοπο ταυτοποίησης, σημειώνω ότι δεν είσαστε υπέρ, αλλά τις τροπολογίες αυτές θα τις συζητήσουμε έτσι κι αλλιώς και αύριο. Φαίνεται λοιπόν ότι θα είναι αποτελεσματικό το αποτέλεσμα με όλα όσα συμπεριλαμβάνει το πακέτο αυτό και αν δεν θέλει κάποιο άλλο το λόγο, Έχουμε εδώ τον κύριο Σέβιντε, ο οποίο είναι ένα τακτικός επισκέπτη τη Επιτροπή μα. και θα θέλαμε να ακούσουμε και τι δικέ σα τοποθετήσεις για τι συμβαστικές τροπολογίε, γιατί βλέπω ότι παρακολουθείτε το θέμα σε όλε τι αρμόδιες επιτροπές. Να σα δώσω λοιπόν το λόγο για να μα πείτε λίγα πράγματα και πώ προχωρούν οι διαπραγματεύσει στο Συμβούλιο για να δούμε αν υπάρχει προπτική συμφωνία σε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ξεκινήσω ευχαριστώντας καταρχάς την εισηγήτρια για την εξαιρετική της δουλειά και τις συμβαστικές τροπολογίες. Οι περισσότερες είναι όντως πολύ καλή συνεισφορά προκειμένου να υπάρξει σύγκληση. Σύγκληση για ένα ικανοποιητικό τελικό κείμενο για το σχέδιο κανονισμού. Έχω μια-δυο επιφυλάξεις βέβαια για αυτά που προτείνονται σε ορισμένες τροπολογίες, συμβαστικέ τροπολογίε, ιδιαίτερω για την πρώτη, την έννοια της παροχής ηλεκτρονικής ταυτοποίησης ω υπηρεσία ε, παροχέα υπηρεσιών εμπιστοσύνης, αυτό δεν συνάδει με τον, με τον ορισμό που περιλαμβάνεται στον κανονισμό έχει. Η παροχή υπηρεσιών ορίζονται βάσει και χαρακτηρίζονται βάσει των υπηρεσιών που παρέχουν. Άρα ε, καθορίζονται από την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και αυτό που σημαίνει ηλεκτρονική ταυτοποίηση. Βέβαια, στην καρδιά της δελειτουργικότητας και της εμπιστοσύνης είναι ακριβώς η προστασία των ηλεκτρονικών συναλλαγών και των σχετικών συστημάτων. Σωστά αναφέρονται λοιπόν αυτά και καλύπτονται και βεβαίως σημεριζόμαστε την πρόθεση να υπάρξει να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα για τα συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Θα πρέπει να είναι ενισχυμένη η ασφάλεια τέτοιων συστημάτων. Πιστεύουμε ωστόσο ότι όλα αυτά μπορούν να γίνουν ακριβώς με ελάχιστες απαιτήσει ασφαλείας. Η έννοια της αμοιβαιότητας όπως έχει συμπεριληφθεί στην τροπολογία υπερθυνοτρία μπορεί παρόλα αυτά να προκαλέσει ένα βαθμό αβεβαιότητας. Γιατί τελικώ μπορεί να είναι αντικείμενο πρόσβαση ή όχι. Ποιο θα είναι το επίπεδο πρόσβαση που θα έχουν δηλαδή οι Ευρωπαίοι πολίτε. Γιατί αυτό, γιατί ο Ευρωπαίο πολίτη που θα πρέπει να γνωρίζει ποιο είναι το σύστημα ταυτοποίηση που έχει κοινοποιηθεί και να γνωρίζεται από τα άλλα κράτη-μέλη, ε, θα πρέπει να το γνωρίζει αυτό. Ιδάλλως δεν θα έχει σαφή εικόνα για το πώ αντιμετωπίζονται τα συστήματα αυτά εκτό τη χώρα του. Τα επίπεδα όμω ασφαλείας μπορεί να μην έχουν συμφωνηθεί βάσει των, ε, του ελάχιστου βαθμού προστασίας. Και θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη η βάση της ταυτοποίησης. Θέλουμε προφανώς να προσφέρουμε κάτι στους Ευρωπαίους πολίτες σε δύο θέσεις. Πρώτα απ' όλα σε ευρωπαϊκό επίπεδο να συμφωνηθούν τα επίπεδα ασφαλείας, αλλά να μην υπάρξει και βεβαιότητα για το τι σημαίνει επίπεδο ασφαλείας, τι μπορεί να είναι αποδεκτό ή όχι βάσει της επιλογής του καθενός από τα συμβαλλόμενα μέρη στα κρατημέλη. Στην ίδια συμβαστική τροπολογία και πάλι έχουμε μια επιφύλαξη για την παράταση της υποχρέωσης ως προς την Ένωση, δεν ξέρουμε αν η νομοθεσία θα διευκολύνει αυτό, η νομική βάση είναι το 149, αλλά αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τουλάχιστον βάση της λειτουργίας των θεσμικών οργάνων μπορεί να λάβει και να αναλάβει δράση διορθωτική για τον κανονισμό που συλλοποιείται από τα κράτη-μέλη. Ε, στην τροπολογία 3 και πάλι, το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας δίνει την εντύπωση ότι η Ένωση, οι φορείς ή τα θεσμικά όργανα της Ένωσης θα βρίσκονται σε θέση να εξοπλιστούν με μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Δεν ξέρουμε αν αυτό θα επιτρέπεται από την συνθήκη όπως ισχύει. Άλλα σημαντικά στοιχεία στα οποία θέλω να σταθώ είναι Εκκοινοποίηση παραβίασης της ασφαλείας. Είναι πολύ σωστό στόχος και το στηρίζουμε διότι προσφέρει διαφάνεια και σαφής, αποσαφηνίζει τις υποχρεώσεις όλων των μερών. Από την άλλη όμως, επιφυλασσόμεθα κάπως για τη συμβαστική τροπολογία, το δεύτερο μέρος της συμβαστικής τροπολογίας, υπάρχουν 7 σε σχέση με την εισαγωγή νέου μέρους αυτού που προσφέρει την ηλεκτρονική ταυτοποίηση στον κανονισμό. Κάτι που δεν είναι αναγκαίο και δεν είναι αντικείμενο του κανονισμού αυτού καθε αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι όσα αναφέρει παράγραφος 2 της συμβαστικής τροπολογίας δεν πρέπει να γίνουν των αντίον, αλλά θα πρέπει αυτό να το επιλύσουν τα κάτι μέλη σε εθνικό επίπεδο, με τις ανάλογες διευθετήσεις και υποχρεώσεις, όπως θα πρέπει να ισχύουν σε κάθε κράτος μέλους. Θα ήθελα επίσης να πω κάτι ως προς τη συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 8. Εκεί υπάρχει το σημείο Β και μια διάταξη που προτείνεται ως προς την αναγνώριση των ε, παροχέων που αναγνωρίζονται διακρατικά και αναγνωρίζονται και από τρίτη χώρα. Είναι σημαντικό σημείο αυτό, γιατί έχει να κάνει και με όσα συμπεριλαμβάνονται στη συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 9. Η η διευκρίνηση αυτή τη διάταξη στην οδηγία θα δώσει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε εγκεκριμένο φορέα υπηρεσιών εμπιστοσύνη ένα κράτο μέλο να μπορεί να ε, εγγυηθεί για έναν άλλον ε, παροχέα τρίτου κράτου. Αλλά πώ θα είναι βέβαιο ότι αυτό ο άλλο παροχέα τη τρίτη χώρα ε, έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία το απαραίτητο επίπεδο και πώς θα διασφαλίσει τα ισοδύναμα μέτρα και την, το επίπεδο προστασία. Το ίδιο και για την ε, διαπίστευση από κάτω μέλος. Μπορεί κάποιος να έχει γκρίνει διαπιστεύσει να σε ένα κάτω μέλος για την παροχή υπηρεσιών που είναι ισοδύναμες με τις υπηρεσίες ε, τις διπηρεσίες, τις ηλεκτρονικές αυτές διπηρεσίες, αλλά και πάλι όταν θα πρόκειται για τρίτη χώρα, πώς θα βαβαιωνόμαστε ότι το επίπεδο ασφαλείας είναι ανάλογο. Δεν μπορούμε να το εγγύθουμε για μια τρίτη χώρα. Βεβαίω, οι αναγνωρίσει αυτέ, αφού λάβουν χώρα, είτε σε επίπεδο των αντικριμένων φορέων ή των κρατών μελών που θα εγγυώνται για τις τρίτες χώρες, όλα τα άλλα κράτη-μέλη θα πρέπει να, ξε... να αποδεχτούν. Θα υπάρχει λοιπόν ε, εξίσωση εδώ με την διαπίστευση και αυτό θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη, ιδίω εάν σκεφτούμε τι στρεβλώσεις μπορεί να προκαλέσουν αυτό το είδους οι αναγνωρίσεις ή διαπιστεύσεις. Τέλος, να ολοκληρώσω με μια σύντομη παρατήρηση για τη συμβαστική παριθμών 14. Εκεί οι φυσικές σφραγίδες και οι ηλεκτρονικές σφραγίδες ε, εξουσιώνονται. Αυτό θα πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε ποια είναι η νομική αξία των ηλεκτρονικών σφραγίδων και να σκεφτούμε τι υποχρεώνουμε τα κράτη-μέλη που χρησιμοποιούν φυσικές φραγίδες ε, να κάνουν. σε κάποιες περιπτώσεις ε, ο ρόλος της φραγίδας είναι πολύ καλά καθορισμένος και αποδεδειγμένα παραδεκτός. Οπότε Σαφώς οι συμβαστικές τροπολογίες είναι μια πολύ καλή συμβολή στην όλη συζήτηση. Τώρα για το πόσο πιθανό είναι να υπάρξει σύγκληση στο Συμβούλιο και πώς προχωρούν εκεί οι διαπραγματεύσεις, αυτά που μπορώ να πω είναι αυτά που και εγώ ίδιος γνωρίζω όμως άμεση αντίδραση. Πολλά σημεία ακόμη συζητώνται στο Συμβούλιο, Ω προς τις συμβαστικές τροπολογίες, βλέπω να υπάρχουν προοπτικές σύγκλησης και για κάποια σημεία στα οποία δεν συμφωνεί απαραίτητα η Επιτροπή, αλλά συνολικά δεν προβλέπουν να υπάρξει κάποια σοβαρή αντίρρηση για να βρεθεί η συμφωνία. Ευχαριστώ. Πολύ μας βοηθήσαν όλα αυτά. Όντως πρέπει να προχωρήσουμε γιατί έχουμε το πακέτο για την ηλεκτρονική ενιαία αγορά. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα το προχωρήσαμε. Τώρα θα δώσω πάλι το λόγο στην ε, Μαρή Καλό για να συνοψίσει. Γιατί έχουμε την ψηφοφορία αύριο, έτσι. Μαρία. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Όπως και εσείς, έτσι και εγώ βρήκα πολύ ενδιαφέρουσες όλες τις παρατηρήσεις σχετικά με τις συμβαστικές τροπολογίες. Εννοείται ότι πρέπει να τις ξαναδούμε λίγο μέχρι αύριο. Πάντως, όπως έχει το πράγμα σήμερα, θα έλεγα ότι η δουλειά έχει γίνει. Για την τελευταία μόνο παρατήρηση όσον αφορά τη διαφορά ανάμεσα στα κράτη-μέλη που έχουν ε, συμβολογραφικές πράξεις και τα λοιπά και εκείνα που δεν έχουν, μα δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία υπόθεση όπου διαπιστώνουμε τέτοιες δυσκολίες. Στη Νομική Επιτροπή ασχολήθηκα με τα κληρονομικά δικαιώματα και να ξέρετε ότι είναι χειρότερα τα πράγματα. Συνεπώς, οι κάποιες δυσκολίες που αναφέρθηκαν διακανονίζονται. Μπορούμε συνεπώς να ψηφίσουμε αύριο βάσει των 14 αυτών συμβιβαστικών τροπολογιών. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Συμμετέχετε και στην Επιτροπή Βιομηχανίας εσείς. Οπότε εκεί μπορείτε να στηρίξετε τα συμφέροντά μας και στον τριμερή διάλογο βέβαια. Στη Ζούρη, όχι στην Ήτρε, διορθώνει η κυρία Γκαλό. Α, ναι, ναι, σωστά. Ναι, μπερδεύτηκα. Ναι, νομικών υποθέσεων, σωστά. Καλώς. Συνεχίζουμε τώρα. Για να δω είναι όλοι εδώ, γιατί έχουμε πάει γρήγορα και δεν ξέρω. Στις 25 λέει το πρόγραμμα ότι πρέπει να αρχίσουμε. Μήπως να σταματήσουμε για 5 λεπτά ή είναι όλοι εδώ. Περιμένουμε κανέναν άλλον. We'll just take a very short break. Θα διακόψουμε για λίγο. Λίγα λεπτά μόνο ώστε να αρχίσουμε στην ώρα μας το επόμενο θέμα. to starting time, hope... Νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε τώρα. Κύριε Μάντερς, έχουμε ακόμα ένα θέμα πριν περάσουμε στο δικό σας. Οπότε βγείτε έξω για το πηγαδάκι σας, αν θέλετε. Η κυρία Ρίγο Πέρες, που είναι συγγήτρια γνωμοδότησης Είναι γνωμοδότηση για ποια επιτροπή, για την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Έχει μεγάλη σημασία όμως για την ενιαία αγορά. Έτσι. Έχουμε ένα σχέδιο γνωμοδότησης, Ιλντίγκο Γκάλ και μετά ε, Κάνεν, σκιώδη συγγήτρια, κύριε Παράνοβα επίσης, θα αντικαταστήσει τον κύριο Βουζό. Δεν ξέρω αν έχουμε εδώ κανέναν από τους πράσινους. Εγώ νομίζω είμαι σκιώδη από τη δικιά μου την ομάδα. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε εδώ κάποιον. Σελήν Τεσβάρτσι; σωστά. Εσείς, μάλιστα. Μετά θα πάρετε εσείς το λόγο. Ίσως αν θέλετε θα μπορούσα να σας παρουσιάσω για το πρόγραμμα δράσης της Επιτροπής. Να ακούσουμε πρώτα την εισηγήτρια και μετά εσείς. Λοιπόν, κυρία Ελντίγκο Γκαλπέλες να μας παρουσιάσει τη γνωμοδότηση. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ξέρουμε ότι η Ευρώπη έχει γεράσει. Που σημαίνει ότι ο πληθυσμός θα συνεχίσει να γυρνάει τα επόμενα χρόνια και άρα θα αυξάνονται οι δαπάνες για την υγεία. Γι' αυτό και χρειάζονται αλλαγές για να διασφαλιστεί η καλή κατάσταση των συστημάτων υγείας. Η υγεία αποτελεί έναν βασικό πυλώνα του κράτους ευημερίας είναι κάτι που το χρειαζόμαστε σε καθημερινή βάση. Η χρήση της όμως και ο τρόπος που εφαρμόζεται αλλάζει. Εξακολουθούν να υπάρχουν μερικά εμπόδια σήμερα τα οποία δεν μας επιτρέπουν να χρησιμοποιήσουμε όπως θα θέλαμε την ε, υγεία. Είτε πρόκειται για τα νομικά πλαίσια τα οποία δεν είναι ικανοποιημένα, ικανοποιητικά είτε πρόκειται για τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε. Η ηλεκτρονική υγεία πάντως θα μπορούσε να βοηθήσει να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής και να βελτιώσουμε την ζωή των πολιτών γενικότερα. Χρησιμοποιώντας καινοτομία. Γι' αυτό πολύ χαιρόμαστε που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παρουσιάσει αυτό το νέο σχέδιο δράσης της προσαρμόζει το παλιότερο προσθέτοντας νέα μέτρα. Ιδιαίτερα βελτιωμένη πρόσβαση στις υπηρεσίε υγείας και περίθαλψης και ισότητα μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών. Επίσης έχει κάνει και μελέτη για τις νομικές πτυχές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας. Πρέπει να επιμείνουμε όμως και σε κάποια ζητήματα τα οποία πιστεύουμε εμείς ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πρώτον, την ανάγκη να υιοθετήσουμε αποτελεσματικά μέτρα στο τομέα της επιστροφής των δαπανών για την υγεία. Ελπίζουμε οι συζητήσεις με τα κράτη-μέλη όσον αφορά τα συστήματα επιστροφής δαπανών για την υγεία θα προχωρήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην εκπλήρωση των προδιαγραφών χρησιμοποιώντας επαγγελματικά στοιχεία κάτι πολύ βασικό για την προστασία των πολιτών. Για την εμπιστοσύνη των ασθενών επίσης, τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας και την σωστή λειτουργία και καλή χρήση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας στον τομέα της υγείας. Δεύτερον, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ούτε όλοι οι πολίτες, ούτε όλοι οι επαγγελματίες του κλάδου είναι εξοικειωμένοι με την χρήση της πληροφορικής. Γι' αυτό θα πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν στη διάθεσή τους μια βοήθεια, μια κατάρτιση κατάλληλα προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους. Τρίτον, είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις την κατάλληλη στήριξη για να έχουν και αυτές πρόσβαση στην αγορά υγείας. Έπειτα να λάβουμε υπόψη μας την ανθρώπινη διάσταση όταν μιλάμε για περίθαλψη ιδιαίτερα όταν μιλάμε για ηλικιωμένους. Τέλος, ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημοσιεύσει ετήσια επισκόπηση της πρόοδου όσον αφορά την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την ηλεκτρονική υγεία στα επιμέρους κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, για το ενδιαφέρον σας και περιμένω τα σχόλιά σας. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών θα είναι 4 Σεπτεμβρίου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Τώρα, οι σκιώδεις εισηγητές πρώτα. Η Αντιπρόεδρος κάνει. Ευχαριστώ πολύ. Αρχίζω με το γεγονός ότι πρόκειται για γνωμοδότηση, που σημαίνει ότι δεν έχουμε αρκετό χώρο βέβαια για να βάλουμε ό,τι θέλουμε. Όμως υπάρχουν κάποια πράγματα που θα ήθελα να υπογραμμίσω και θα ήθελα να συμπεριληφθούν και στην ηλεκτρονική υγεία και στη γνωμοδότησή μας. Από πού έρχονται τα χρήματα για να προωθηθούν οι πρωτοβουλίες για τις πλατφόρμες για την ηλεκτρονική υγεία. Ελπίζω να μπορούμε να πούμε ότι η ηλεκτρονική υγεία θα μπορέσει να αποτελέσει μέρος της εμβληματική πρωτοβουλίας ε, για, για τη στρατηγική μας για το 2020. Να συμπεριλάβουμε δηλαδή το θέμα της γύρανσης του πληθυσμού. Δεύτερον, θα ήθελα να δω και τα τρία διαφορετικά επίπεδα της ηλεκτρονικής υγείας. Εννοείται ότι είναι πολύ σημαντικό οι ειδικοί, οι εμπειρογνώμονες να συμπεριληφθούν ένας γιατρός δηλαδή που ειδικεύεται στην ηλεκτρονική υγεία, εννοείται ότι θα έπρεπε να τον ρωτήσουμε αν είναι ειδικό ακόμα και αν δεν είναι γιατρός δηλαδή. Και τους πελάτες φυσικά, τους ασθενείς. Όταν πρόκειται για EGD, όταν πρόκειται για ακτινοβολία. οι γιατροί, οι ασθενείς θα πρέπει να πούνε την γνώμη τους. Έχουμε ένα καλό σύστημα νοσοκόμων όμως. Πρέπει να αναπτυχθεί περισσότερο το θέμα των ε, φαρμακοποιών, γιατί οι φαρμακοποιοί και οι νοσοκόμοι είναι ο ενδιάμεσος κρίκος ανάμεσα στον ασθενή και τον γιατρό. Γνωρίζουμε ότι οι ηλικιωμένοι πρέπει να παίρνουν ε, την φαρμακευτική τους θεραπεία όσο γίνεται πιο γρήγορα, αλλά μερικές φορές καθυστερούν γιατί δεν έχουν τη συνταγή. Ενώ αν κάποιος νοσοκόμος μπορεί να πάει σπίτι, ελέγξει την κατάσταση, τι έχει και τι δεν έχει από φάρμακο ασθενής και μέσω της ηλεκτρονικής υγείας συμβουλευτεί το γιατρό, τότε θα μπορούσε πολύ πιο γρήγορα να ε, πει στον ασθενή τι αντιβιωτικά ή τι άλλα φάρμακα θα έπρεπε να πάρει. Έτσι λοιπόν η ηλεκτρονική υγεία μπορεί να βοηθήσει περισσότερο τους ηλικιωμένους αλλά ακόμα και όσους ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Κάτι άλλο που λείπει από την πρωτοβουλία αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι προτάσεις σχετικά με τις δυνατότητες που έχει ο ίδιος ασθενής. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση και να ακουστεί η φωνή του ασθενή περισσότερο. Με την κατάλληλη κατάρτιση μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να ασχοληθούν οι ίδιοι με την ε, υγεία τους και να μπορούν μέσω του προγράμματος ηλεκτρονικής υγείας να απευθυνθούν οι ίδιοι στους γιατρούς. Θα έπρεπε και αυτό να το δούμε παραπέρα. Και θα μπορούσαμε βέβαια και να επενδύσουμε να δέρχομαι στον ορίζοντα 2020 να βρούμε ένα σύστημα που να ελέγχει την κατάσταση υγείας των ασθενών και να το έχουν ε, οι άνθρωποι να συνδέονται με αυτό και έτσι να πηγαίνουν τα αποτελέσματα στις ιατρικές υπηρεσίες. Τέλος. Θα ήθελα πιο συγκεκριμένες προτάσεις για τη γνωμοδότηση αυτή και για το πρόγραμμα ηλεκτρονικής υγείας. Ξέρω βέβαια πώς είναι δύσκολο. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα, αν μη τι άλλο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει πώς θα αντιμετωπίσει το θέμα της διαλειτουργικότητας των διαφόρων συστημάτων που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη σε μία χώρα, με μια μεγάλη χώρα, είναι δύσκολο, πόσο μάλλον μεταξύ πολλών και διαφορετικών χωρών φιλοδοξίες είναι μεγάλες. Αν μη τι άλλο, τα συστήματά μας θα έπρεπε μεταξύ τους να είναι συμβατά. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Η τοπαϊκή από την Επιτροπή. Κύριε Πάνομα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστή. Συγγνώμη. Κύριε Πάνομα, είναι πάρα πολύ δύσκολο το θέμα αυτό και είναι πολύ δύσκολο να έχουμε μια καλή ποιότητα γνωμοδότηση στο περιορισμένο πλαίσιο που προδιαγράφεται. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να πω ότι τα πιο πολλά θέματα καλύπτονται από την προτινόμενη γνωμοδότηση. Θα ήθελα να αναφέρω κανένα δύο θέματα. Το θέμα δεν είναι μόνο η βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών στην υγειονομική περιθάλψη με τα μέτρα περικοπών ε, που γίνονται σχεδόν σε όλα τα κρατημέλη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και ουσιώδες και αναπόφευκτο για τα κρατημέλη να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές για την διαχείριση των οικονομικών πόρων και τη βελτίωση παρόλα αυτά της πρόσβασης. Δεν είναι εύκολο αυτό και γι' αυτό λοιπόν θα μπορούσε να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση το e-health, η ηλεκτρονική υγεία, όχι μόνο για τη διαχείριση των ε, νοσημάτων, αλλά και για τη διαχείριση των βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των νοσοκομείων, μεταξύ των σχετικών εμπλεκομένων αρχών. Το Θέμα επίσης που τίθεται αφορά την επαγγελματική κινητικότητα. Αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση σε παγκόσμιο επίπεδο. Ιδιαίτερα για τα κράτη-μέλη εκείνα τα οποία ουσιαστικά παρέχουν τους επαγγελματίες στον τομέα της υγείας σε άλλα κράτη-μέλη. Και σε αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει η ηλεκτρονική υγεία, το e-health, αλλά φυσικά εδώ τίθεται και το θέμα της ευθύνης. Όταν παρέχονται τέτοιες υπηρεσίες, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου γίνονται εξετάσεις από αλλοδαπούς ιατρούς στην επικράτεια ενός κρατός μέλους ενό κράτου σε ασθενή από τρίτο κράτο μέλο. Ε, σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν πάρα, πολλές, ε, πολλά προβλήματα και περιπλοκές. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει κάποιες ε, προτάσεις και ενδεχόμενες επενδύσεις που θα μπορούσαν να επιλύσουν τα θέματα αυτά. Για το θέμα της ικανής χρήσης των τεχνολογίας πληροφοριών και της ικανής αξιολόγησης των θέματων υγείας. Κοιτάξτε, όλοι υποθέτω αφότου έχουν βγάλει την ιατρική, έχουν κάποιες βασικές γνώσεις ε, σε τεχνολογίες πληροφοριών, αλλά και πάλι δεν επαρκεί αυτό. Μιλάμε για πολύ ψηλό επίπεδο εφαρμογών και για μια σειρά προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν για την ασφάλεια του ασθενή και μιλώντας για την ασφάλεια του ασθενή και για θέματα ευθύνης για, σε περίπτωση παροχής ηλεκτρονικής ε, υγείας, τίθεται το θέμα και της προστασίας των δεδομένων. Αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί. Και θα πρέπει προφανώς να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή σε αυτό το θέμα. Τέλος, κλείνοντας, να μιλήσω για την αγορά μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όχι μόνο στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, αλλά και στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών. Μέχρι σήμερα, τεράστια, τεράστιος όγκος μικρομεσαίων επιχειρήσεων που εργάζονται για την παροχή νέων λύσεων ε, ηλεκτρονικής υγείας, διαπιστώνουν ότι τα συστήματα αυτά δεν είναι διαλειτουργικά, δεν είναι σημαντικά τα μέντα δε θα χρειαστεί κατά πάσα πιθανότητα πολύ μεγαλύτερη συνεργασία και καθοδήγηση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι επιχειρήσει αυτέ που θέλουν να παρέχουν τέτοια προϊόντα στην αγορά, προκειμένου να διασφαλιστεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο για την ασφάλεια του ασθενή. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρο. Η κυρία Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω και πάλι την κυρία Παραναβά για τον τρόπο με τον οποίο μιλάει και θεωρώ ότι όπως πάντα μας έδωσε μια καλή επισκόπηση της κατάστασης. Ένα θέμα θα ήθελα να υπογραμμέσω, το θέμα του empowerment, των ικανοτήτων του ίδιου του ασθενή. Στην Ήπεθρο άτομα μεγαλύτερης ηλικία, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτά τα άτομα να ξεπεράσουν το ψηφιακό χάσμα. Γιατί, ξέρετε, με τις περικοπές ουσιαστικά υπονομεύονται εκείνοι τους οποίους πρέπει να βοηθήσουμε πιο πολύ από κάθε άλλον. Πώς μπορούμε λοιπόν να φροντίσουμε αυτό το ψηφιακό χάσμα να μην πλήξει τους ε, πιο ηλικιωμένους. Κάποια σημεία και από την ομάδα μου λέει ο Πρόεδρος. Νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση προσθέτουμε ε, επιπρόσθετα στοιχεία στο έργο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. Αυτό που μου προκάλεσε έκπληξη είναι ότι περιλαμβάνονται πολλά στοιχεία για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την αίσθηση ότι είναι υποαναπτυγμένες ε, οι διαστάσεις ε, του IT, της ε, τεχνολογίας πληροφοριών και ξέρουμε, για παράδειγμα, πόσο περίπλοκη είναι η ανάθεση συμβάσεων για ξενοσοκομεία, τι πολιτικέ προκλήσεις ενέχονται και νομίζω ότι οι συνάδελφοι το γνωρίζουν. Τι θα πω. Θα πρέπει να κοιτάξουμε και θέματα δημοσίων συμβάσεων σε ό,τι αφορά τις καινοτομίες στον ιατρικό κλάδο, γιατί Μιλάμε για ένα κλάδο όπου μπορούν τα θέματα ηλεκτρονικής υγείας να συνεργαστούν με τα νοσοκομεία για την πρόταση πιλωτικών προγραμμάτων. Και με χαρά μου θα υποβάλλω τέτοιες τροπολογίες προς την εισηγήτρια. Γιατί Είμαστε σε φάση τελικής διατύπωσης των κειμένων με το Συμβούλιο, αλλά θεωρώ ότι είναι σημαντικά τα ζητήματα αυτά. Αυτό αφενός. Κατά δεύτερον, νομίζω ότι σε ό,τι αφορά θέματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης, είναι πολύ σημαντική η διάσταση αυτή και όπως είπατε και εσείς κύριε Ρούλε, σε πολλές περιπτώσεις έχουμε απέναντί μας ηλικιωμένους ασθενείς. Μιλάμε λοιπόν για την ασημένια οικονομία. Είναι ένας νέος όρος αυτός που αναφέρεται. Αλλά αφετέρου, θεωρώ Δεν ξέρουμε λοιπόν τι θα γίνει στο μέλλον σε ό,τι αφορά την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης. Ίσως όμως θα έπρεπε να γίνει εκπαίδευση και άλλων ατόμων. Δεδομένης όμως και της ε, ανεργίας μεταξύ των νέων, θα πρέπει να δούμε και τις σχετικές επενδύσεις που γίνονται για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Και αυτό το έφτασε την προηγούμενη πέμπτη στη συζήτησή μας. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τα άτομα τα οποία μπορούν να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν επαρκώς τις τεχνολογίες αυτές και θεωρώ λοιπόν ότι μία από τις βασικές μας επενδύσεις στην καταπολέμηση της αλλεργίας των νέων είναι ακριβώς η ανάπτυξη τέτοιων ικανοτήτων και αν θέλετε μετά η ανάπτυξη ενός στρατού νέων οι οποίοι θα μπορούσαν να εφαρμόσουν αυτά τα συστήματα και να εξηγήσουν στον ασθενή πώς μπορούν να χρησιμοποιεί τα νέα αυτά εργαλεία. Εκπαίδευση λοιπόν ε, των νέων, αλλά προώθηση τελικά και της ε, υγείας. Τελευταίο ε, ζήτημα, το οποίο καλύπτεται, έχει να κάνει με την προστασία των δεδομένων. Νομίζω ότι στον τομέα της υγείας εν γέννη απόλυτα σαφές πλέον και υπήρχαν πολλές ε, δημοσιεύσεις σε ό,τι αφορά βάσεις δεδομένων και ε, υγειονομική περίθαλψη. Προφανώς είναι, έχουν υποστεί μια διαδικασία ανωνυμοποίησης ε, τα στοιχεία αυτά, αλλά η αντίδραση ό,τι αφορά τον καρκίνο, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ε, όπου πολλές περιπλοκές παρουσιάζονται και υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ των ασθενών και υπάρχουν πάρα πολλές εκδοχές καρκίνου. Για να μπορέσουμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε σε ευρία κλίμακα την ε, ανταπόκριση στην θεραπεία θα βοηθήσει γενικότερα στην καλύτερη αντιμετώπιση της ασθένειας. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιούνται αυτά τα στοιχεία πάντα ε, με το άρο ότι γίνεται σεβαστή, σεβαστό το απόρτο του ασθενή. Εκφράστηκαν ανησυχίε για τα ιδρύματα, τα ερευνητικά, για κάποια από τα στοιχεία του πακέτου για την προστασία δεδομένων που ενδεχομένω να παρεμποδίσουν τα στοιχεία αυτά. Θα πρέπει λοιπόν στην Επιτροπή μα να το κοιτάξουμε αυτό. Αυτά λοιπόν από δική μου πλευρά. Κανεί άλλο από την Επιτροπή θέλει να πάρει το λόγο. Έχετε το λόγο, κυρία Να προσθέσω κάτι. Μετά από όλη τη συζήτηση που κάναμε, νομίζω ότι η προστασία των δεδομένων είναι ζωτική σημασία εδώ. Μιλάμε για έναν τομέα ε, γοργά αναπτυσσόμενο και μιλάμε για δεδομένα ευαίσθητα, γενετικά δεδομένα, ακόμα και για το γονότυπο. Είναι σημαντικό λοιπόν ποιος έχει πρόσβαση και τι μπορεί να ανακύψει να το λάβουμε υπόψη. Um, Άρα, να καλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την κυρία Ταβάτσε, εάν προφράσω στο το όνομά σα, να μας δώσει τη δική της άποψη και μετά θα δώσω το λόγο στην κυρία Ριγκόνη Πέρες να συνοψίσει. Ευχαριστώ. Θα ακολουθήσω λίγο πολύ τα σχόλια που έλαβα, πρώτα απ' όλα από την εισηγήτρια. Υπογραμμίζει την ανάγκη τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν στην εναρμόνιση της, των επιστροφών σε σχέση με την ηλεκτρονική υγεία, το e-health. Έχουν, έχουν ξεκινήσει σχετικά οι συζητήσεις με τα κράτη-μέλη. Το ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη εκπαίδευση των πολιτών και των επαγγελματιών του χορηγίας. Για τους πολίτες το θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς το έχετε επισημάνει και εσείς για τους πιο ηλικιωμένους και εδώ η ενεργός γύρανση και σχετική πρωτοβουλία και τελική σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ σημαντική για να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ε, δραστήρια άνθρωποι την άποψη της του, του χρονικού διαστήματος που παραμένουν ενεργοί. Ω προ την προστασία δεδομένων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι και αυτό είναι θεμελιώδε, μια και έχουμε να κάνουμε με ιατρικά δεδομένα. Αλλά σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε τώρα, πρέπει να περιμένουμε πρώτα απ' όλα το σχέδιο κανονισμού να εγκριθεί, να γίνουν συζητήσει και να ολοκληρωθούν και μετά θα σχολιάσουμε για το αποτέλεσμα της έρευνας, της συγκατάθεσης. Για την ώρα είμαστε στα χέρια σας. Και άλλη μια παρατήρηση για την ε, ανάληψη της ευθύνης από τους ασθενείς. Εδώ να τονίσω ότι Αυτό στο δίσιο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν ένας από τους βασικούς μας στόχους, μια από τις δράσεις που προβλεπόταν και στην ψηφιακή ατζέντα της Ευρώπης. Οι ασθενείς να έχουν πρόσβαση στους ε, διάφορους κωδικούς και σε αυτό το της του 2015, αλλά στα πλαίσια του ορίζοντα 2020 προσπαθήσαμε να συμπεριλάβουμε στους μελλοντικού μας σκοπούς και διαφορετικές πηγές σηματοδότησης για να αναλάβουν την ευθύνη τους οι ασθενείς με πιο αποτελεσματικό τρόπο και για τη διαλειτουργικότητα όπως θα δείτε και στο πρόγραμμα δράσης είναι ένα από τα πρώτα μας μελήματα υπάρχουν εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διαλειτουργικότητα αλλά να τονίσω απλώς το εξής για να τονωθεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων κρατών μελών υπάρχει και το δίκτυο του e-health, της ηλεκτρονικής ε, υγείας που δημιουργήθηκε βάσει τη οδηγία για τα δικαιώματα των ασθενών και το δίκτυο αυτό λειτουργεί και ασχολείται με τη διαλειτουργικότητα ανταλλαγή δεδομένων για τα ιατρικά ε, αρχεία τα ιστορικά των ασθενών. Θέλει να ορίσει ένα σύνολο πληροφοριών που θα είναι ουσιαστικά το ιστορικό, το βιογραφικό ενό ασθενού. Στόχο είναι να έχει κανεί ε, σύνοψη των ιατρικών πληροφοριών, να ανταλλάσσονται εύκολα, κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε και βεβαίω θα διευκολύνει πάρα πολύ την κινητικότητα των ασθενών στην Ευρώπη. Θα βοηθήσει όμω και τα κράτη-μέλη, διότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν προβλήματα με την εφαρμογή των ρητρών για την ηλεκτρονική υγεία. Εάν λοιπόν υπήρχε διαλειτουργικότητα έστω και για τη μορφή, το έντυπο, τις πληροφορίες που θα λαμβάνουν οι γιατροί όταν κανείς ταξιδεύει στους ασθενείς, θα ήταν πολύ εξυπηρετικό αυτό. Και στο δίκτυο έχουμε ακολουθήσει τα πορίσματα του πολύ χρήσιμου πολιτικού προγραμμάτος της ΕΠΣΟ με τις ιατρικές πληροφορίες, την σημασιολογία, και τα αρχεία των ασθενών. Προκειμένου να υπάρχει διαλειτουργικότητα μεταξύ κατώμελων, θα πρέπει κανεί να μπορεί να μεταφράσει έναν ιατρικό όρο, μια ιατρική έννοια από τη μια χώρα στην άλλη. Αυτά χάρη στην έψω έχουν ε, προχωρήσει. Το, το, ο χώρο τη ηλεκτρονική υγεία είναι ένα τομέα, που υπάρχει ανταλλαγή βελτιστών πρακτικών μεταξύ κρατών μελών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβάλλει εδώ. Και με αυτό το στόχο κατά νου χρηματοδοτήσαμε το σχετικό, ευρωπαϊκό, ευρωπαϊκό ιστότοπο που καλύπτει και πολλά άλλα ζητήματα και την ηλεκτρονική υγεία. As uh, the comment you've made on that I... Για τι τεχνολογίε επικοινωνία και πληροφορία, όντω δεν έχουν αξιοποιηθεί αρκετά στον τομέα τη υγεία, μα δίνουν τεράστιο δυναμικό και θα συμφωνήσουμε, έχουμε μια καθυστέρηση εδώ, πρέπει να την καλύψουμε. Ένας από τους βασικούς λόγους για αυτή την καθυστέρηση είναι το θέμα της εμπιστοσύνης. Η υλοποίηση της ηλεκτρονικής υγείας στα κάτι μέλη πολλές φορές δημιουργεί δυσκολίες διαλειτουργικότητα. Και αυτό όντως πρέπει να το μελετήσουμε, την εμπιστοσύνη των πολιτών με συγκεκριμένες προτάσεις και λύσεις, αλλά και την εμπιστοσύνη των επαγγελματιών που φοβούνται Πρέπει κανείς να εγγυηθεί την ασφάλεια, οπότε μια από τις δράσεις μας, μέσα από το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, είναι να σκεφτούμε το θέμα της έννοιας της εμπιστοσύνης. Μια πράσινη βίβλος για την ηλεκτρονική υγεία και το πώς την αντιλαμβανόμαστε. Κάτι που θα ετοιμαστεί το 2013, τον Οκτώβριο του 2013. Ευρύτερες διαβουλεύσεις με όλους τους ενδιαφερομένους στην Ευρώπη και τις εφαρμογές στον τομέα της υγείας. Οι εφαρμογέ αυτές έχουν τη δυνατότητα να διευκολύνουν τα κράτη-μέλη στην εξοικονόμηση πόρων και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων. Αυτή τη στιγμή ίσω όλα αυτά να μην είναι ασφαλή, να μην συναντούν πλήρω με την νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό ξεκινήσαμε τι ευρύτερε διαβουλεύσει για να κάνουμε ό,τι μπορούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να βελτιώσουμε την ασφάλεια, τη διθεσιμότητα των ηλεκτρονικών τύπων και την ε, συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα το απόγευμα και ευχαριστούμε που μας ενημερώσατε. Είναι ένα σημαντικό θέμα. Κύριε Ρικό η σειρά σας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως είπε και η κυρία Πέτικανεν, πέρα από το ότι πρέπει να είναι περιορισμένη η γνωμοδότηση αυτή, τα σχόλιά σας βοηθούν να τις δώσουμε μεγαλύτερη πυγμή. Υπάρχουν διάφορα θέματα που ακούστηκαν και πιστεύω και εγώ ότι είναι πολύ σημαντικά. Ξεκινάμε πράγματι από διαφορετικά συστήματα υγείας στις διάφορες χώρες μέλη. Το σύστημα δημόσιας υγείας στη χώρα μου, για παράδειγμα, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε εξαιρετικό. γιατί χρησιμοποιεί την πληροφορική, την επικοινωνία για να εκδημοκρατιστεί ακριβώς το σύστημα αυτό και για να μπορούμε να έχουμε στη διάθεσή μας τους καλύτερους ειδικού. Άκουσα και τα σχόλια της κυρίας Παρανόβα για τις βέλτιστες πρακτικές και την ανταλλαγή αναφέρθηκε στην ασθένεια. Πράγματι, όλες οι τεχνολογίες πληροφορικής πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι κάτι βασικό και οι ασθενείς θα πρέπει να δίνουν τη συγκατάθεσή τους για να μπορεί κανείς να τα χρησιμοποιήσει. Άρα οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν περισσότερες δυνατότητες να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο σύστημα ηλεκτρονικής υγείας για να μπορούν ακριβώς να έχουν ε, υγεία. Μπορούμε επίσης εδώ να λάβουμε υπόψη μας και τους νέους, ιδίως εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου πολλοί νέοι είναι στην ανεργία. Οι νέοι λοιπόν θα μπορούσαν να συμμετάσχουν και να βοηθούν τους ηλικιωμένου να κατανοήσουν πράγματα τα οποία τους είναι πάρα πολύ δύσκολα, πληροφορική δηλαδή. Κατά τα σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τα σχόλιά σας. Το θέμα της ε, κυβερνοϊγείας είναι ένα θέμα που βέβαια μας απασχολεί όλους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι πράγματι 4η Σεπτεμβρίου. Οπότε στις διακοπές σας, ε, στην παραλία να σκέφτεστε και τι τροπολογίες θέλετε να υποβάλλετε. 24 Σεπτεμβρίου θα τις εξετάσουμε, 30 Σεπτεμβρίου θα ψηφίσουμε και τον Οκτώβριο θα πάει στην Ολομέλεια. Καλώς, περνάμε τώρα στο τελευταίο μας θέμα για σήμερα. Είναι του Τόιν Μάντερς. Πρόκειται για νομοθετική έκθεση σχετικά με την απλοποίηση της μεταφοράς μηχανοκίνητων οχημάτων ταξινομημένων σε άλλο κράτος εντός της ενίας αγοράς. Τι χρειαζόμαστε πράγματι την απλοποίηση. Υπάρχουν 27 συμβαστικές τροπολογίες που θα πρέπει να εξετάσουμε πριν ψηφίσουμε αύριο. Γι' αυτό το ΕΝΜΑΝΤΕΣ θα πρέπει να μας τις παρουσιάσει. Το ΕΛΚΕΚ προσωπείται εδώ. Α, ήρθε ο κύριο Κάρα, Α, δεν σας χαρεί. Συγγνώμη, γλιστρήσατε εδώ, μπήκατε στην αίθουσα, δεν σα πηρίλησε. Είναι εδώ λοιπόν ο κύριο Κάρα, η κυρία και η Διαρούλα και εγώ είμαι εδώ. Οπότε για πρώτη φορά σήμερα θα έλεγα ότι έχουμε full house εδώ. Α το γιορτάσουμε. Και α αρχίσουμε με τον κύριο Μάντερς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Και το Ποσίκα που βοήθησε τόσο πολύ. Ευχαριστώ τους κοιόδες εισηγητές, γιατί πάντα γίνονται αλλαγές της τελευταίας στιγμής. Αλλά εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Τι προσπαθούμε να πετύχουμε λοιπόν εδώ προσπαθούμε να καταλήξουμε σε συμβαστικές λύσεις για τα πιο σημαντικά θέματα τα οποία θέτουν οι πολιτικές ομάδες. Τώρα αναφερόμαστε στα επιχειρήματα, γιατί μπορεί να αρνηθεί μια χώρα ένα όχημα. Για παράδειγμα, εάν δεν υπάρχει ασφάλεια αστικής ευθύνης. Υπάρχει δηλαδή κατάλογος πια σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να αρνηθεί μια χώρα. Ή ότι οι πολίτες δεν μπορούν δύο φορές να διξονομήσουν το όχημά τους. Αναφερόμαστε και στις κυρώσεις αν κάποιος δεν έχει ταξινομήσει το όχημά του έγκαιρα. Υπάρχουν αυτά στις συμβαστικές προτάσεις. Νομίζω ότι έχουμε βρει κοινό τόπο αν χρησιμοποιείται πάνω από 6 μήνες σε μια χώρα το όχημα, τότε πρέπει να υπάρξει κάποια ενέργεια από τον ιδιοκτήτη. Όπως επίσης το θέμα της αμοιβαίας αναγνώρισης της ταξινόμησης ήταν πολύ σημαντικό και για τον κύριο Καρά ότι μια τέτοια ταξινόμηση μπορεί να χρησιμοποιεί, να χρησιμεύσει και διασυνοριακά. την ε, μηδέα αναγνώριση επίσης των ε, οδικών ελέγχων. Γιατί την ταξινόμηση είναι πολύ σημαντικό. Γιατί μπορεί να ελεγχθεί μια εβδομάδα ένα όχημα και μετά πάτε στην νέα σας χώρα και ελέγχεστε και εκεί. Ε, δεν είναι καλό αυτό, δεν αρέσει βέβαια στον κόσμο. είναι μια από τις μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες από ό,τι λένε. Και βάζουμε και κάποιες ρήτρες ασφάλειας κατά των απατών. Το θέμα της φορολογίας δηλαδή, ότι η χώρα ταξινόμησης έχει δικαίωμα να ζητήσει το φόρο. Υπάρχει ένα software που χρησιμοποιούν πολλές χώρες όπου συνδέονται βάσεις δεδομένων οι εθνικές μεταξύ τους. Και έτσι θα υπάρχει μια ευρωπαϊκή, εικονική ευρωπαϊκή βάση δεδομένων. Και γιατί την ευρωπαϊκή, γιατί θα είναι διάφορες εθνικές οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους. 27 συμβαστικές τροπολογίες έχουμε. σε μία θα αναφερθώ που είναι αριθμός 23, είναι της τελευταίας στιγμής. Στην πρώτη παράγραφο λέμε πιο θετικά το ίδιο πράγμα. Το διατυπώνουμε θετικά. Και λέμε όπου συνάδει με το τη ρύθμιση της χώρας ε, μέλος μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τα χρώματα της Ένωσης. Ελπίζω να το υπερψηφίσετε αύριο. Έχουμε και κάποιες επιπλέον αιτιολογικές σκέψεις για να εξηγήσουμε γιατί εισάγουμε διάφορα πράγματα και γιατί η νομική βάση έχει ως έχει. Τώρα θέλω να ακούσω τα σχόλια των συναδέρφων. Ας αρχίσουμε τον κύριο Κάρα τότε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη συνεργασία μεταξύ των ε, βοηθών και του εισηγητή ήταν πραγματικά εξαιρετική. Νομίζω ότι καταλήξαμε σε ένα καλό συμβιβασμό και ο συμβιβασμό περιλαμβάνει de facto 10 βασικές ε, αξιώσεις. Στην τελευταία, στην τελευταία διατύπωση, σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά χρώματα στις πινακίδες, πρέπει να σας πω ότι Είναι σημαντικό να περάσουμε από την αρνητική σε μια θετική διατύπωση. Γι' αυτό αποτελεί το στόχο για την ενιαία αγορά. Κάθε πινακίδα είναι, αν θέλετε, και μια κάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν να το πάρουμε πολύ στα σοβαρά το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ποιος είναι ο επόμενος. Κυρία Στάιλερ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον εισηγητή, να τον ευχαριστήσω για όλη τη δουλειά που έκανε και για τις συμβαστικές τροπολογίες. Από πλευράς της ομάδας μας, ε, μας ε, χαροποιεί η συμπερίληψη της αστικής ευθύνης, αν και θα, προσπα... θα προτιμούσαμε όλα τα οχήματα να είναι ασφαλισμένα πριν μπουν στους δρόμους. Καλωσορίζουμε παρ' αυτά την προσθήκη του στοιχείου αυτού. Έχουμε ανησυχίες για την τροπολογία 27 που ζητά εφαρμογή μετά από τρία έτη. Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ίσως θα μπορούσαμε να βρούμε μία μέση λύση. Να ορίσουμε δύο έτη ως ε, μία ενδιάμεση λύση. Να δω και τι λένε οι συνάδελφοι. Είναι σημαντικές λοιπόν και 26 συμβαστικές τροπολογίες. Ε, νομίζω λοιπόν ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει μια ε, ενιαία διαμόρφωση όλων των προδιαγραφών προκειμένου να καταπολεμηθεί και το διασυνοριακό έγκλημα. Σας ευχαριστώ και πάλι συγητά και όλες τις ομάδες για τη συνεργασία τους και προσβλέπουμε στην αυριανή ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ρούλα. Ναι, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πολύ καλή συνεργασία, για την μεγάλη διάθεση σύναψης συμβιβασμών. Πραγματικά σας ευχαριστώ και ελπίζω αύριο να καταλήξουμε στο ευκταίο αποτέλεσμα. Να γίνουν αποδεχτές ε, οι συμβαστικές τροπολογίες, γιατί ασφαλώς το επόμενο βήμα είναι οι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο. Και αυτό θα πρέπει να μα απασχολεί να ολοκληρώσουμε την έκθεση αυτή στην τρέχουσα θετία Είναι τεχνικό το ζήτημα. Λίγα είναι δηλαδή ουσιαστικά τα θέματα στα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε διαφωνία με το Συμβούλιο και είναι σημαντικό λοιπόν να περάσουν τα θέματα αυτά. Και αν για παράδειγμα ο κ. όπως εγώ δεν θα είναι στην επόμενη θετία εκ των πραγμάτων, είναι σημαντικό να ολοκληρωθούν τώρα τα ζητήματα αυτά. So um, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, και εγώ θα είμαι από τα μέλη που δεν θα συμμετέχουν στις ευρωεκλογέ. Να σας πω το εξής. Στου τομείς, στους τομείς στους οποίους επικεντρώνεται η έκθεση αυτή. Απλοποίηση. Απλοποίηση της μεταφοράς των οχημάτων Νομίζω ότι οι πιο πολλές διατάξεις σχετίζονται με το θέμα αυτό και ο εισηγητής έχει κάνει σπουδαία δουλειά. Συμφωνούμε από αυτού. Και συμφωνούμε επί των ε, συμβιβαστικών τροπολογιών. Να τονίσω αυτό που είπε και η κυρία Ρούιλε, πόσο, πόσο σημαντικό είναι να περάσει γρήγορα η έκθεση αυτή. Ο Τουάν Μάντερς πραγματικά είναι εξαιρετικός σε ό,τι αφορά την ε, διεύρυνση των προτάσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με κάθε δημιουργικό τρόπο. Και θυμάμαι ε, τις ετικέτες, για παράδειγμα, για τα κλωστοϊφαντουργικά προϊόντα που καταφέραμε να συμπεριλάβουμε ένα σωρό προτάσεις για το πώς θα πρέπει να πλένονται τα ρούχα κτλ. Σε ό,τι αφορά επίσης ε, μια άλλη οδηγία, καταλήξαμε να τον εξαναγκάσουμε να ε, αποσύρει κάποιες από τις προτάσεις του, οι οποίες δεν ήταν καθόλου, δεν μπορούσαμε καθόλου να τις δικαιολογήσουμε. Αν περάσει όμως η νομοθεσία αυτή, θα αλλάξει ο τρόπος καταχώρησης των οχημάτων και το κατά πόσο θα υπάρχουν συστήματα GPS ε, μέσα στις πινακίδες των οχημάτων, πρέπει να σας πω ότι αυτό δεν έχει να κάνει τίποτα με το πεδίο εφαρμογής του, της έκθεσης. Ε, δεν απλοποιεί καθόλου την διαδικασία. Για πινακίδες που βρίσκονται σε διαμετακόμιση, θα χρειαζόταν συσκευή ραδιοταυτοποίησης. Αυτό θα σημαίνει μια ολόκληρη ε, επένδυση, νέες ναι, συσκευές, δεν υπάρχει καμία σχετική ανάλυση, δεν υπάρχει καμία σχετική προδιαγραφή και συνάδελφοι εγώ συστήνω να το απορρίψουμε αυτό ως πρόταση γιατί αν θέλουμε να το εξετάσουμε, να το εξετάσουμε αλλά ξεχωριστά και επίσης με ανησυχεί και αυτή η πρόταση για κοινέ πινακίδε, τη χρήση τη Ευρωπαϊκή Σημαία κτλ. Και πάλι αυτό δεν εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογή ε, του νομοθετήματο. Αν θέλουμε να περιπλέξουμε το να περάσει το, η πρόταση αυτή από το Συμβούλιο, τι να πω. Πολύ συναρπαστικέ ιδέε αυτέ του Τουάν Μάντερ και είναι γενικά καλό το ρόλο του Άι Βασίλη και κρεμάει όλο και πιο πολλά τώρα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρώ όμω ότι θα πρέπει να απορριφθούν. Αν θέλουμε να κάνουμε μια ξεχωριστή έκθεση, να την κάνουμε για τα θέματα αυτά. Αλλά πιστεύω και σα το υπενθυμίζω συνάδελφοι ότι η πρόταση αυτή είναι απάντηση σε συγκεκριμένε καταγγελίε των πολιτών. Και οι πολιτέ δεν ανησυχούν για τι πινακίδε και το χρώμα του και για το κατά πόσον έχουν σύστημα ραδιοσυχνική ε, ταυτοποίησης. Όχι. Το πρόβλημά τους είναι το πόσο αργή είναι η διαδικασία καταχώρησης, μεταφοράς κτλ. Ας επικεντρωθούμε λοιπόν σε αυτά αύριο. Να ψηφίσουμε αυτά αύριο, να ξεκινήσουμε την διαπραγματεύση με το Συμβούλιο, να δούμε πώς μπορούμε να υποφελήσουμε τους πολίτες, γιατί αν ε, προσθέσουμε όλα τα υπόλοιπα στοιχεία, θεωρώ ότι θα περιπλέξουμε περιτά την όλη διαδικασία. Η ε, κυρία Γκέπχαρτ έχει το λόγο. Κυρία Γκέπχαρτ, έχει το λόγο. Κανείς άλλος. Uh, ε, Η ε, κυρία Γκέπχαρτ. Νομίζω ότι ο κύριος Μάντερς έχει πάντα καλές ιδέες, αλλά συμφωνώ μαζί σας. Βασικά εδώ πέρα έχουμε κληθεί να ανταποκριθούμε στις ανησυχίες του πολίτη. Και ήταν λοιπόν ένα πάρα πολύ σημαντικό αίτημα αυτό του πολίτη, ότι θα πρέπει να απλοποιηθεί η διαδικασία μεταφοράς ενός οχήματος και καταχώρησης ενός οχήματος. Αν ε, προσθεθούν οποιαδήποτε προβλήματα, είτε λόγω άδεια, είτε λόγω ασφάλειας, είτε λόγω ε, τεχνικού ελέγχου, είτε λόγω κακής συνεννόησης μεταξύ των κρατών και αυτό θεωρώ ότι είναι το χειρότερο. Σε αυτά λοιπόν καλούμαστε να απαντήσουμε, προκειμένου οι πολίτες να δουν και κάτι θετικό από την Ευρώπη. Νομίζω ότι σε αυτά θα πρέπει να επικεντρωθούμε. Σε αυτά θα πρέπει να ρίξουμε το βάρος μας. Αλλά να προτείνω στον κύριο Μάντερς να κάνουμε μια προφορική και γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να θέσουμε τα άλλα θέματα. Νομίζω όμως ότι σωστά τα λέτε Πρόεδρε, θα πρέπει να φροντίσουμε να μην την παραφορτώσουμε την πρόταση αυτή και προκειμένου να μην διακινδυνεύσουμε να μην κάνουν τελικά τίποτα τα κρατημέλη σε ένα θέμα που πραγματικά πρέπει να συμβούν κάποιες αλλαγές. Ο κύριος Κάρας, λέει ο Πρόεδρο, κανεί άλλο. Ο κύριο Κάρα. Καταρχά, νομίζω θα πρέπει να κοιτάξουμε τη θετική διάσταση, τα 10 αυτά ζητήματα που αφορούν την απλοποίηση, την απλοποίηση των διαδικασιών για τον πολίτη στην ενιαία αγορά. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα, σε αυτό συμφωνούμε όλοι, de facto. Κατά δεύτερον, το θέμα των πινακίδων. Εδώ είναι μια μακρά διαδικασία είναι της σημασία. Και προτείναμε να το κοιτάξουμε και σε μία μελέτη αντικτύπου. Να ζητήσουμε μία έρευνα μία μελέτη, γιατί εμείς απλά θέλουμε να ενισχύσουμε και να συνεχίσουμε την διαδικασία αυτή είναι μια μελέτη αντικτύπου. Αν θα μπορούσαμε με τη μελέτη αντικτύπου αυτή να αναφέρουμε και να προωθήσουμε στο επόμενο βήμα την σκέψη αυτή, το υποστηρίζουμε. Υποστηρίζουμε την εξέλιξη αυτή. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει σαφής διάκριση των ε, θεμάτων αυτών. Να ορίσουμε ποια είναι τα πιο σημαντικά και ποια είναι τα τρεβούσια σημασία. Ο Πρόεδρος. Θέλετε να ακούσετε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κύριε Μάντερς, πριν ξαναπάρτε το λόγο. Θα μπορούσατε να μας ε, κάνετε κάποιες προτάσεις για το πώς να αντιμετωπίσουμε και τις πολύ δημιουργικές ιδέες, δεν λέω, του κύριου Μάντερς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και καλησπέρα σας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τις θέσεις της για τις τροπολογίες που προτάθηκαν στις 27 Ιουνίου. Νομίζω λοιπόν ότι στην συνάντηση τότε σημειώσαμε ότι όντως για τα επιπρόσθετα αυτά στοιχεία που περιέχονται στην πρόταση Μάντερς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι ακόμα σε θέση να παρουσιάσει τη θέση της καθότι δεν περιλαμβάνοντας στην αρχική πρόταση για το θέμα της ε, ραδιοτεχνικής ε, ταυτοποίησης, για το θέμα των πινακίδων. Όλα αυτά δεν αποτέλεσαν ε, αντικείμενο της πρότασης και γι' αυτό λοιπόν δεν υπάρχει σχετική μελέτη. Άρα όντως ναι, δεν συμπεριλαμβανόντουσαν στην αρχική πρόταση. Κατανοούμε το στόχο. Συμφωνούμε και με την, με την ιδέα της διεύρυνσης, αν θέλετε, του αισθήματο του ευρωπαϊκού. Ενοποιώντας ε, τα χρώματα και την όψη των πινακίδων. Αλλά και πάλι. Επαναλαμβάνω ότι δεν τα έχουμε μελετήσει αυτά και την πρότασή μας. Όπως ε, προαπαιτείται, με μελέτες αντικτύπου κτλ. Τώρα, για τη συζήτηση. δεν μας ενημέρωσαν για τις ε, σε μεμβαστικές τροπολογίες. Από ό,τι ακούω από τη συζήτηση, χαιρόμαστε που έχει προχωρήσει η ιδέα για την αμοιβαία αναγνώριση των πινακίδων και των ελέγχων, των τεχνικών ελέγχων. Αλλά προκειμένου να σας παρουσιάσουμε την οριστική μας θέση, θα πρέπει να δούμε και τις τροπολογίες, τις οποίες ακόμα επαναλαμβάνω δεν τις έχουμε δει. Αυτά λοιπόν από δική μου πλευρά. Σας ευχαριστούμε. Ο Τουάν Μάντερς. Θέλετε να συνοψίσετε. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Κοινοβούλιο και οι πολιτικοί γενικώ τείνουν να προσθέτουν πράγματα σε ένα θέμα. Μετά συζητάνε, αλλά έχουν ρόλο και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ. Α συντηρήσουμε ο καθένα λοιπόν την αρμοδιότητά του και α μην τα μπλέκουμε πριν φτάσουμε στο Συμβούλιο. Θα υπάρξουν και διαφωνίε. Νομίζω όμω οι πρωταρχικοί στόχοι όπω του προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλύπτονται. Καλύπτονται Λάβαμε πάντως πολλά σχόλια για το σύστημα ταξινόμησης. Στη Γερμανία ήδη εφαρμόζεται σε ένα βαθμό και είναι πολλοί οι πολίτες που φοβούνται να αγοράσουν όχημα σε άλλη χώρα διότι δεν ξέρουν αν έχει κλαπεί ή όχι. Πρέπει να τους βοηθήσουμε. Πρέπει να βελτιώσουμε την εύρυθμη λειτουργία της ε, ενιαίας αγοράς με μια ενιαία πινακίδα. Έτσι οι πολίτες δεν θα χρειάζεται να μπαίνουν σε νομικές ε, ατραπούς. Θέλουμε να βελτιωθεί λοιπόν η λειτουργία της ενιαίας αγοράς και μιλάμε για δύο με 4 αυτοκίνητα, ε, ευρώ ένα όχημα. Άρα είναι πολλά και χρειάζεται μελέτη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι να πω. Συμφωνήσαμε στι συμβαστικέ τροπολογίες και αύριο υποθέτω ότι θα εγκριθεί η 23η συμβαστική τροπολογία και ελπίζω ότι οι συνάδελφοι συντονιστές θα συμφωνήσουν. Χρειαζόμαστε μελέτη αντικτύπου Εάν είναι πολύ αρνητική τοποθέτηση, όπως μπορούμε να φανταστούμε, τα ξανασυζητάμε. Αλλά τώρα πρέπει να ψηφίσουμε, γιατί ήθελε να αναβληθεί ψηφοφορία, αλλά μου είπανε όχι, όχι. Είναι μία από τις μεγαλύτερες πηγές σύγχυσης για όλους, αν δεν περάσει αυτό, οπότε ας ψηφίσουμε και ας συγκριθεί και μελέτη αντικτύπου, εφόσον χρειάζεται. Πάντως, σίγουρα πρόκειται για μεγάλη βελτίωση της εκ νέου ταξινόμησης και οι νομικές υπηρεσίες καλύπτονται. Αυτά. Ελπίζω αύριο ψηφοφορία να πάει καλά. Θα δούμε το αποτέλεσμα όμως. Είμαι πολύ θετικός και αισιόδοξο και ελπίζω ότι εν τέλει Λόγω χάρη δίνουμε και σε εσά τρία χρόνια περιθώριο για την ε, μεταφορά. Ζητάτε βέβαια να μειωθεί. Δεν ξέρω πώ μπορείτε να αλλάξετε τη συμβιβαστική. Μπορείτε αύριο να υποβάλλετε προφορική τροπολογία για τα τρία ή δύο έτη. Αλλά δική σα είναι η τροπολογία, εσεί θα κάνετε ό,τι θέλετε. Εμεί συμφωνήσαμε στα δύο. Εάν ακολουθήσετε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πάρουμε τώρα ένα χρόνο. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε πολιτικοί, για να αφήνουμε περιθώριο στις κυβερνήσει και να βελτιώνουμε τη ζωή των πολιτών. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Α ψηφίσουμε αύριο. Και όλοι νομίζω με καλή συνεργασία θα καταφέρουμε να συμβάλλουμε στο αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Όλοι το ίδιο είπατε. Θα ψηφίσουμε αύριο και θα συζητήσουμε το τι έγινε. Το πρόβλημα με την πρότασή σας είναι το θέμα της αναλυτικότητας. Το μόνο που μας απασχολεί εδώ είναι η εκ νέου ταξινόμηση. Εάν μιλάμε για ευρύτερα ωφέλη για τους πολίτες, το θέμα είναι αν θα πρέπει να αλλάξει το σύστημα ταξινόμησης και των πινακίδων για όλα τα οχήματα ή αν είναι πολλά αυτά τα οχήματα που θα ταξινομούνται εκ νέου. Βάσει της πρότασής σας, μόνο τα οχήματα που είναι ταξινομημένα σε μια χώρα θα καλύπτονται. Ο στόχο δεν είναι να αλλάξει το σύστημα ταξινόμηση στα κράτη-μέλη. Τουναντίον, αντίον, μόνο η επαναταξινόμηση μα ενδιαφέρει. Εσεί τι λέτε, να αλλάξουν εκ βάθρων τα συστήματα ταξινόμησης. Εάν δουλεύει το σύστημα και έχουμε πολλές επαναταξινομήσεις, δίκιο έχετε. Το σύστημα μέχρι τώρα δουλεύει και η Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων, όπως προτείνουμε, θα μπορούσε να δημιουργηθεί και τα κάτι μέλη θα είναι ελεύθερα. Θα είναι ελεύθερα να το εισάγουν είτε με το δικό τους εθνικό σύστημα ταξινόμησης, είτε όχι. Είναι ένα πρώτο βήμα μόνον. Δεν είναι ένα ταξίδι στο φεγγάρι. Ταξινόμηση οχημάτων είναι, αλλά μπορεί να είναι ένα μεγάλο άλμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεκινήσουμε με αυτό το μικρό βήμα και αν δούμε ότι λειτουργεί, τα κράτη-μέλη θα λάβουν τα μέτρα του. Αν μπλοκάρουμε όμω τι βελτιώσει και τι εμποδίζουμε, ε, τι θα γίνει, δεν θα γίνει τίποτα στο τέλος. Ε, χρειάζεται καινοτομία, χρειάζεται κοινοτόμο σκέψη. Τη στιγμή που η οικονομία δεν τα πάει καλά γιατί οι πολιτικοί δεν μετακινούνται, δεν θέλουν να καινοτομήσουν, δεν θέλουν να αλλάξουν το μέλλον, αυτό είναι συντηρητισμός μετά. Γι' αυτό είμαστε πολιτικοί, για να είμαστε φάνταστοι, να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και να έχουν εμπιστοσύνη στο μέλλον τους οι πολίτες, με καινοτομία. Ωραία. Πολύ φιλοσοφική τοποθέτηση. Ας δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Σίγουρα στους πολίτες θέλουμε να δείξουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε αποτελέσματα και θα πρέπει βεβαίως να συμφωνήσουν 28 κράτη-μέλη πολύ γρήγορα αν θέλουμε να προχωρήσει καιρός για τις εκλογέ. Δεν είμαι βέβαιος ότι η φιλοσοφία της κοινοτομίας, της πινακίδας των οχημάτων θα αλλάξει την πορεία του κόσμου όπως λέμε στα αγγλικά. Δεν ξέρω αν θα χαθεί και κάποιο φορολογικό εισόδημα όπως ε, σήμανε οι συνάδελφοι. Ίσως να μην υπάρξει καθολική συμφωνία με τις ιδέες σας κύριε Μάντερς. Μας απασχολούν και άλλα πρακτικά ζητήματα, αλλά τέλος πάντων. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε. Okay. Well, thank you very much. Well, we're going to be a... Ευχαριστούμε πολύ. Θα ψηφίσουμε αύριο και θα μπορούν όλοι να εκφραστούν για τις προτάσεις του κυρίου Μάντερς. Και μετά θα δούμε αν θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει με τα κράτη-μέλη. Ξέρω ότι η Λιθουανική Προεδρία ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το θέμα. Ωραία. Να σα ευχαριστήσω όλου και να σα θυμίσω ότι η συνεδρία μα αρχίζει αύριο στι 9. Εδώ. Για μια σημαντική συζήτηση για την ε, ε, ε, ενιαία πολιτική. Θα ψηφίσουμε βέβαια και μην ξεχάσετε τι κάρτε σα. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Κυρία Γκέπχαρτ, θα χρειαστεί να με βοηθήσετε για το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα πωλήσεων. Και εσείς κύριε Μάιντερ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.